Να ξεκινήσουμε με 10 λεπτά καθυστέρηση. Παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα καταρχάς, εξ ονόματος όλων των συναδέλφων της Επιτροπής Αλίας, να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας οι οποίοι έχουν έρθει για να παραστούν σε αυτή την ακρόαση με αντικείμενο τις γυναίκες και τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, στις ζώνες αλίας η κυρία Επίτροπος θα έρθει αλλά με λίγη καθυστέρηση και έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί μας για να μας πει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα σας δώσω το λόγο και όταν έρθει η κυρία Επίτροπος θα ολοκληρώσει ο μιλητής ο εκάστοτε. Στο τέλος της ομιλίας του θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να κάνει τη δική της παρέμβαση. Καλώς ήλθατε λοιπόν και πάλι. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγνώμη για την ισχνή παρουσία συναδέλφων σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Ωστόσο, πολλές άλλες επιτροπές αυτή τη στιγμή συνεδριάζουν. Όσοι είμαστε παρόντες θελήσαμε να έρθουμε εδώ, όσοι είναι παρόντες δεν μου έχουν ανακοινώσει το λόγο της απουσίας τους. Επομένως δεν μπορώ να σας πω περισσότερα από αυτό. Βλέπω ότι έχουμε ισχυρή γυναικεία αντιπροσώπευση και ίσως αυτό είναι καλό, γιατί θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά ε, για τα θέματα αυτά. Γνωρίζουμε ήδη ως Επιτροπή κάποιους από τους προσκεκλημένους μας. Άλλους τους συναντήσαμε στο πρόσφατο σεμινάριο που είχε διοργανώσει ε, η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή. Νομίζω ότι όλοι οι προσκεκλημένοι έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στην κυρία Αντρές Παρέα, υπεύθυνη, αρμόδια για την πολιτική που αφορά στην ισότητα των ευκαιριών. Γεια σας. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, καλώς ήλθατε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Αντρές Βαρέα και αμέσως μετά, ε, εάν συμφωνείτε κυρία Δαμανάκη, να δώσω σε εσάς το λόγο. Επομένως πρώτα η κυρία Βαρέα και μετά η αξιότιμη κυρία Επίτροπος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κυρία Επίτροπε στην Επιτροπή μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους αλλά και όλους τους παριστάμενους σε αυτή την ακρόαση. Είναι σαφές ότι σήμερα ε, είναι ισχνή η παρουσία των μελών της Επιτροπής Αλίας, διότι και άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου συνεδριάζουν σε διπλανές αίθουσες και πολύ συχνά αυτό δυσκολεύει τις εργασίες μας και αφαιρεί από τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε τη λάμψη τους. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, που η Επιτροπή ασχολείται με το ρόλο των γυναικών σε σχέση και με την αλληλεία. Αυτή η ανάγκη φάνηκε και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο κατάρτισης και υιοθέτησης διαφόρων εκθέσεων. Μιλούμε επίσης για το ρόλο της γυναίκας στην βιώσιμη ανάπτυξη στις ζώνες αλίας. Έχουμε την έκθεση Πατράου της ε, συναδέλφου. Κάθεται εξ αριστερών μου και εκεί σε αυτή την έκθεση ένα άρθρο ε, αναφερόταν στη γυναίκα συγκεκριμένα. Πάντοτε ο τομέας αυτός ήταν σημαντικός. Ωστόσο, η, κοινωνία έχει δώσει ένα ρόλο στη γυναίκα, ο οποίος δεν έχει φανεί σε όλες του τις διαστάσεις. Μιλούμε για την ηχθειοκαλλιέργεια, για την μεταποίηση, για τη θέση σε εμπορία, αλλά και για την, ε, τις συμπληρωματικές οικονομικές δραστηριότητες. Ο ρόλος της γυναίκας λοιπόν δεν έχει φανεί ξεκάθαρα. Ε, λόγω της ε, διαίρεσης των φύλων και των διαφορών δεν έχει φανεί ο ρόλος της γυναίκας. Παραδοσιακά θα έλεγα ότι οι γυναίκες ασχολούνταν περισσότερο με την καλλιέργεια της γης και οι άντρες περισσότερο με την αλλιευτική δραστηριότητα στην θάλασσα. 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν αλλιευτική δραστηριότητα και ως προς την ε, ως προς την αλία, ε, το 4,19% διενεργείται από γυναίκες. 6% στην Ελλάδα, λίγο αυξημένο το ποσοστό στην Ιταλία και στην Πορτογαλία 14% οι γυναίκες. αλλά και στο μεταποιητικό κλάδο ως προς την ελευτική δραστηριότητα η γυναίκα διδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το 75% των εργαζομένων είναι γυναίκες σε αυτό τον κλάδο και 25% μόνο άνδρες. Θα μπορούσα να σας δώσω και παραδείγματα αναζώνες και περιοχές. Στη Βαλτική, για παράδειγμα, 17.480 γυναίκες. Κατά πλειοψηφία λοιπόν οι γυναίκες στο κλάδο αυτό. Στη Γεωργία οι γυναίκες ε, αντιστοιχούν στο 47,1%. Πλησιάζουμε δηλαδή το 50%. Εδώ λοιπόν ο τομέας που μας ενδιαφέρει έχει πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Οι γυναίκες μπορούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά και υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Διάφορες επαγγελματικές διέξοδοι ανοίγονται και θα μπορούσαν οι γυναίκες να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ειδικά σε τομείς και σε περιοχές όπου ε, υπάρχει πρόβλημα με τις καινούργιες γενιές και είναι δύσκολο να φανεί ποιος θα πάρει τη σκητάλη στο μέλλον. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα από την Ισπανία. Έχουμε στην Παγιόν ή στην ευρύτερη περιοχή της Γαλλικίας ενώσεις που έχουν λάβει επαγγελματικό χαρακτήρα και θέλουν ουσιαστικά να καταπολεμήσουν τη μαύρη εργασία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι γυναίκες συνήθως κάνουν δουλειές χωρίς πολλά, που δεν απαιτούν πολλά προσόντα και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων. Για το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας θέλει να ενισχύσει την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και να στηρίξει τις εθνικές και τοπικές οργανώσεις και ενώσεις. Δύο είναι οι άξονες προτεραιότητες. Ε, ο τέταρτος άξονας είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η βιώσιμη ανάπτυξη των αλληλευτικών ζωνών, αλλά και η ενθάρρυνση ε, μέσων δημοσίου συμφέροντος μέσω από τις ε, συλλογικότητες τις διάφορες. Θα πρέπει να δουλέψουμε ώστε τα επόμενα χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υιοθετηθεί η σωστή στρατηγική και η διάσταση του φύλου να μπει σε όλες τις κοινοτικέ πολιτικές. Η γυναική απασχόληση να αυξηθεί, οι μισθοί να εξισωθούν, οι γυναίκες να αντιπροσωπευθούν καλύτερα στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αυτές είναι οι γραμμές τις οποίες θα πρέπει να τονίσουμε, να υπογραμμίζουμε συνεχώς όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας θα πρέπει να λειτουργήσει και για να προστατεύσει την ισότητα των ευκαιριών. Επικροτούμε τη σύσταση, τη δημιουργία ισπανικού δικτύου ε, ενώσεων γυναικών που δραστηριοποιούνται στον αλλιευτικό τομέα. Ελπίζουμε αυτό να γίνει και σε άλλες χώρες, ώστε ε, στο μέλλον να καταλήξουμε σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μια ευρωπαϊκή οργάνωση. Υπό αυτή την έννοια είναι ενδιαφέρον να ε, προβάλλουμε και να προάγουμε την αμοιβαία ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση μεταξύ των διαφόρων φορέων και γυναικείων οργανώσεων. Να γίνει ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών, ώστε να ενταχθεί καλύτερα η γυναίκα στον τομέα της αλίας, αυτό τον αλληλευτικό κλάδο γενικότερα θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο η θέση της γυναίκας σε αυτόν τον κλάδο και να εξετάσουμε καλύτερα τις πολιτικές που έχουμε θεσπίσει. Να υπενθυμίσω επίσης ότι ε, και σε εθνικό κρατικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, έχει καθιερωθεί και κατοχυρωθεί νομικά η ισότητα των φύλων. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Άρα καλό θα ήταν να ενημερώνονται καλύτερα ε, τα διάφορα όργανα που συμμετέχουν στην εκάστοτε διαβούλευση. Η, εργασία σε δίκτυο, όλη αυτή η δικτύωση μεταξύ των ενώσεων και οργανώσεων είναι κάτι το πολύ θετικό, διότι μόνο έτσι προκύπτουν οι βέλτιστες πρακτικές. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να στηρίξουν όλες αυτές τις προσπάθειες, κυρίως να έρθουν να καλύψουν το κενό που δημιουργείται με την έλλειψη πόρων απότερος στόχος είναι η ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στον αλλιευτικό κλάδο. Έχουμε τις ε, γυναίκες που ε, ε, ασχολούνται με την καλλιέργεια οστρακοειδών στη Γαλλικία ή γυναίκες που ασχολούνται με την αλληλεία στην Βαλένθια, την περιοχή από την οποία προέρχομαι εγώ, κατάγομαι εγώ. Βεβαίως μένει να καλύψουμε πολύ μεγάλη απόσταση για να φτάσουμε στην πραγματική ισότητα και να ε, δουλέψουν για αυτή όλες οι επίσημες αρχές. Στόχος είναι να φανεί με πιο ορατό τρόπο η θέση της γυναίκας στον κλάδο της ώστε να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στις ζώνες αυτές και ελπίζουμε, ελπίζω πραγματικά η σημερινή ακρόαση να λειτουργήσει ε, ως ένα φόρουμ από το οποίο θα προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις εργασίας, συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα για να βελτιωθεί η θέση της γυναίκας. Ε, τίποτα άλλο κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια θα συμπεριλάβουμε τα συμπεράσματα ε, των επόμενων ομιλητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια έχω την τιμή να σας παρουσιάσω την Επίτροπο για την Αλία και τις θαλάσσιες δραστηριότητες, την κυρία Δαμανάκη, που θα σας προσφωνήσει και έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα των γυναικών στην Αλία. Έχετε, καλώς ήρθατε κυρία Δαμανάκη, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητές κυρίες ε, και αγαπητοί κύριοι, σπάνιοι κύριοι που είναι εδώ παρόντες. Ο κύριος Γκάλαχαρ είναι πάντοτε μια εξαίρεση, ε, είναι το μόνο ε, μέλος άνδρας της Επιτροπής που είναι εδώ παρόν. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ε, την πληροφορία ότι η Κομισιόν υιοθέτησε την χάρτα για τις γυναίκες για την πρόθεση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς πολιτικής το Σεπτέμβριο εφέτος. Πριν από δύο μήνες η Κομισιόν υιοθέτησε μια περιεκτική στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την υλοποίηση των στόχων της χάρτας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιστεύω ότι σήμερα αυτή η ακρόαση είναι, έρχεται εν ευθέτω χρόνο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη και συνάδει ε, με τις ε, πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα και όλη την Επιτροπή για την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και θα ήθελα επίσης να τους ευχαριστήσω που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστώ σχετικά με το θέμα αυτό γενικά. Η υποχρεωσή μου, πρόθεσή μου είναι να βεβαιωθώ ότι οι αρχές ε, της χάρτας ε, θα καλύπτουν, θα ε, περάσουν σε όλο τον τομέα της αρμοδιότητάς μας. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου όσον αφορά και την αλληλεία και τις θαλάσσιες ναυτιλιακές υποθέσεις. Τώρα όμως θα εστιαστώ στην αλία, διότι η ακρόαση σημερινή αφορά την αλία. Η προώθηση της ισότητας των γυναικών στον τομέα αυτό δεν είναι μόνο ε, θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι κάτι το απαραίτητο για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο στις παράκτιες περιοχές και για να επιτύχουμε ε, το στόχο μιας ανάπτυξης ε, ε, που πλήρους ε, που θα περιλαμβάνει όλους μέχρι το έτος 2020. Συμφωνώ με κυρία Αντρέας Μπαρέα. Θα σας μιλήσω εν συντομία για ε, τα δύο θέματα θα ήθελα να μιλήσω σήμερα για τον ρόλο των σημερινών των γυναικών στην αλληλεία και κυρίως στην βιώσιμη ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη της αιλιάς και μετά θα περάσω στις δράσεις που προγραμματίζουμε για το προσεχές μέλλον, ώστε να δώσουμε πρωτεύοντα ρόλο στις γυναίκες στην πολιτική μας. Οι γυναίκες ακούσαμε τους αριθμούς στα στοιχεία, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι γυναίκες ήδη παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από 100.000 ε, γυναίκες απασχολούνται στον τομέα της αλίας, δηλαδή εν τέταρτο ε, του ενεργού δυναμικού του τομέα. Αυτή η σημασία βεβαίως ε, ποικίλει ανάλογα με τους υποτομείς. 4% στον τομέα της αλίας, αλλά στις υδατοκαλλιέργειες ε, έχουμε 39% γυναίκες και στο μεταπητικό τομέα έχουμε 56% γυναίκες. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτυγχάνουν ε, να αναγνωρίσουν έναν ορισμένο αριθμό σημαντικών παραγόντων. Τα στοιχεία δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας πω μερικά πράγματα περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολλές γυναίκες είναι αόρατες στις στατιστικές, δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση. Έχουμε αυτό το ε, κοινό φαινόμενο αλλά δεν ε, απασχολούνται επίσημα ε, και δεν επωφελούνται από την κοινωνική ασφάλιση, για να μην αναφέρουμε με μερικές από τις γυναίκες που επισκευάζουν τα δίκτυα, τα μπαλώνουν ή που μαζεύουν κοχύλια και όστρακα και που δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτό που δεν μας λένε τα στοιχεία είναι ότι πολύ συχνά ε, ε, ε, οι γυναίκες έχουν επίπονες εργασίες και η συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για την διαχείριση των πόρων ή τα δικαιώματα, τα αλλιευτικά, η συμμετοχή τους είναι πάρα πολύ περιορισμένη στη λήψη αποφάσεων. Τα στοιχεία δεν δείχνουν την σημαντική ε, συμβολή ε, στον κοινωνικό ιστό των τοπικών αλλιευτικών κοινοτήτων. Αυτό το τελευταίο σημείο έχει μεγάλη ε, σχέση με τη σημερινή συζήτηση, γι' αυτό θα επεκταθώ. Μιλήσαμε για την έξυπνη ανάπτυξη και την καινοτομία. Στην Αλία θα βρείτε ότι οι γυναίκες πάρα πολύ συχνά διαφοροποιούνται και προσθέτουν αξία, προστιθέμενη αξία στις κοινότητές τους, διότι βρίσκουν ε, νέους τρόπους μεταποίησης και εμπορίας ασχολούνται με εναλλακτικούς τομείς που έχουν σχέση με τα ψάρια, με την αηλία. Ε, δηλαδή κυρίες, ε, οι κυρίες, ε, οι γυναίκες καινοτομούν. Καινοτομούν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα ε, τέτοιων έξυπνων πρωτοβουλειών ε, των γυναικών. Γυναίκες ε, που αναπτύσσουν μικρές μονάδες μεταπητικές για τελικά προϊόντα υψηλής, υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητας που πολλούνται σε ακριβές τιμές ή βρίσκουν άμεσα τρόπους πώλησης και κρατούν τα ψάρια, το προϊόν μέσα στην κοινότητα. Έχουν ε, επίσης εστιατόρια, εστιατόρια ε, ψαριών. Επίσης οργανώνουν επισκέψεις σε διάφορες μονάδες. Πριν από δύο εβδομάδες στην διάσκεψη CFCP της ε, διάσκεψης. Είχαμε αυτή τη διάσκεψη για την μεταρρύθμιση, ήταν προκαταρκτική, προπαρασκευαστική. Μάθαμε ε, για μια ομάδα γυναικών στην Γαλλική που αποφάσισαν να κάνουν κάτι ε, για την κακή ποιότητα των αποθεμάτων. Οι δύο γυναίκες παρουσίασαν ε, την πρωτοβουλία του όπου οι συλλέκτες που σπάρνακα έχουν να κάνουν αυτά τα μειονεκτήματα μέρα με τη μέρα για να βρούνε έναν τρόπο ρύθμισης και ελέγχου της ε, τιμής αγοράς ε, των μαλακίων αυτών και των μηδιών. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα καινοτομικής πρωτοβουλίας γυναικών και θα ήθελα να τις ευχαριστήσω που το κάνουν αυτό. Ε, αυτά τα σχέδια μικρής κλίμακος και υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι αυτό που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε ε, στο μέλλον. Ε, Χάρη involved into local βεβαίως έχουμε συμπράξεις, συνεργασίες σύμφωνα ε, με μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω. Μπορούν επίσης ε, να έχουν χρηματοδότηση για να αρχίσουν επιχειρήσεις σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός, ε, τα τρόφιμα ή η ανανεώσιμη ενέργεια. Εναλλακτικά, οι γυναίκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια για να βαθμίσουν ε, τα προσόντα, την εξειδίκευση για προσαρμοστικότητα, για πρόσβαση στην απασχόληση, κυρίως προς όφελος των γυναικών. Αργότερα σήμερα το απόγευμα η Μόνικα Μπέρτ από την Μονάδα Υποστήριξης ε, του ε, Δικτύου Αλίας, Φέρνε όπως την ονομάζουμε, θα σας παρουσιάσει τις δυνατότητες που, η που προσφέρεται για πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ισότητα με τον φίλων είναι ε, μια από τις πρωτεύουσες, πρωταρχικές αρχές ε, του Ταμείου Αλίας θα πρέπει να υποστηριχθούν σχέδια και προγράμματα που ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα της αλίας και στην ανάπτυξη των αλλιευτικών κοινοτήτων. Εκτός από την πρόσβαση στα κονδύλια υπάρχει επίσης και υποστήριξη για μέτρα κοινού συμφέροντος όπως η δικτύωση, η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των οργανώσεων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών όπως επίσης και συνειδητοποίηση. Αυτά για την κατάσταση σήμερα. Θα σταματήσω εδώ και θα, σταθώ, θα στραφώ στο μέλλον και πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, την έλλειψη ορατότητας και αναγνώρισης για τις γυναίκες, ούτως ώστε να οικοδομηθεί ο ρόλος τους στον τομέα της αλίας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ε, την δημιουργία ε, γυναικείων οργανώσεων σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό. Και ε, θα πρέπει βεβαίως ε, να προωθήσουμε την ανάπτυξη την παράκτεια. Η Ισπανία είναι ένα καλό ε, παράδειγμα που έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα γυναικών. Ο κύριος Θεράνο θα μας μιλήσει γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα των Ισπανών. Θα ήθελα να ακολουθηθεί το παράδειγμα το ισπανικό και να δημιουργηθούν δίκτυα αλλού. Όταν λειτουργήσουν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γενικών, ε, γυναικών ούτως ώστε να, υπάρξουν, να υπάρξει ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, περισσότερη ορατότητα για τις γυναίκες και αναγνώριση, να γίνουν περισσότερο γνωστές. Δεν δεν πρέπει να έχουμε αποτελέσματα ε, και στοιχεία βεβαίως. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη αξιολογούν ε, την υλοποίηση των κονδυλίων, την χρησιμοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Ταμείου. Ε, πόσα κονδύλια δόθηκαν απευθείας σε γυναίκες, μέχρι ποιου βαθμού το Ταμείο χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση των ίσων ευκαιριών. Η αξιολογήση που θα γίνει τον Ιούνιο 2011 θα μας πει ε, τι έγινε έχω ήδη ζητήσει από τις υπηρεσίες μου να γίνει αυτή η αξιολόγηση από τα αποτελέσματα. Θα αντλήσουμε διδάγματα για το πώς θα μπορούμε να αυξήσουμε το mainstreaming ε, μεταξύ για να ληφθεί δηλαδή υπόψη ισότητα των φίλων στην πολιτική μας. Θα έχουμε μια νέα μελέτη για τον ρόλο των γυναικών ε, στον ε, τομέα της αλίας και την ανάπτυξη των παρακτήων περιοχών. Από τα αποτελέσματα θα έχουμε την βάση για μια διάσκεψη το δεύτερο εξάμεινο του 2011. Αυτή η εκδήλωση θα παράσχει επίσης μια πλατφόρμα για να συζητηθούν εμπειρίες και να διερευνηθεί ε, πώς ε, τα άτυπα δίκτυα ε, σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όπως το ακτέα θα μπορούν να έχουν περισσότερη σημασία. Η ακτέα επίσης θα κάνει μια παρουσίαση εδώ σήμερα από ό,τι ξέρω. Επίσης, θα προωθήσω την δημιουργία παρομοίων ε, δικτύων στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας. Εάν ε, δοθούν οι ευκαιρίες οι γυναίκες ε, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια μας. Θα πρέπει να τους δώσουμε την δυνατότητα. Αν τους δώσουμε την δυνατότητα, την ευκαιρία, θα υποφεληθούν. Θέλουμε να βασιστούμε σε αυτό εφ' και ε, να αντλήσουμε από τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι γυναίκες για να απτύξουν ε, τις δυνατότητες ε, των αλλιευτικών περιοχών. Θα πρέπει οι γυναίκες να αντιπροσωπεύονται σε όλα τα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια. Δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη, αλλά έχουμε ήδη λάβει μέτρα. Έχουμε ε, εμπλέξει την, ε, τις γυναίκες στον προβληματισμό μας για την μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, συμμετοχή στις ε, διαβουλεύσεις όπως αυτή που έλαβε χώρα πριν από δύο εβδομάδες. Οι υπηρεσίες μου εξετάζουν τώρα την δυνατότητα οργάνωσης ειδικών εργαστηρίων για τον ρόλο των γυναικών στην αλία και εξετάζουμε τρόπους ε, για να προωθήσουμε ε, τα καλύτερα προγράμματα, σχέδια και πρωτοβουλίες γυναικών. Έχουμε την μονάδα Farnet. Αυτή η μονάδα έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη τα θέματα ισότητας των φύλων για την διαφοροποίηση και την τοπική διακυβέρνηση. Υπάρχει ήδη μια ομάδα ε, εργασίας στο Web Forum είναι ένας χώρος για δικτύωση, για ανταλλαγή μεταξύ πρωταγωνιστών, μεταξύ ε, γυναικών και για την βιώσιμη ανάπτυξη των ηλιευτικών περιοχών. Η ακτέα ε, το δίκτυο οργανώσεων γυναικών στην Αλληλεία και την Ιδατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη παίζει σημαντικό ρόλο. Ε, για να κλείσω κυρίες και κύριοι, έχουμε περισσότερους κύριους τώρα. Ε, η ανάγκη να ενισχύσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην Αλία είναι σημαντική. Εργάζονται σκληρά και υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ρόλο τους στην ε, Αλία και την προστιθέμενη αξία που παράγουν και υπάρχει ε, μεγάλη απόσταση με, το, με την ε, κοινωνική αναγνώριση της οποίας την χάνουν. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα. Ως γυναίκα και ως επίτροπος πρέπει λοιπόν να μην φυστώ καμιάς προσπάθειας για να διορθάσω αυτή την ανισορροπία. Η ε, μελλοντική μεταρρύθμιση μας δίνει μια καλή ευκαιρία να το πράξουμε αυτό. Όπως γνωρίζετε, προγραμματίζουμε μεταξύ άλλων την αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων και για τα άτομα που δουλεύουν στον τομέα. Και αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, να αυτονομήσουμε τις γυναίκες, να τους ενισχύσουμε την αυτονομία τους. Ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε για τα λόγια σας, στην προσφώνησή σας. Ελπίζουμε ότι τα άκουσαν με μέγιστη προσοχή αυτές τις καλές προθέσεις ε, που έχετε για το έργο που θα αναπτύξετε στο μέλλον όσον αφορά τις γυναίκες στην Αλία. Και εφ' θα περάσουμε τώρα κιόλας στο πρώτο μέρος της ακροάσεως που αφιερώνεται στα δίκτυα και σε ενώσεις γυναικών στην Αλία. Θα δώσω σε κάθε μια από τις γυναίκες που θα παρεύουν 8 λεπτά μέγιστο χρόνο ώστε να μπορέσουμε μετά να έχουμε μια συζήτηση πρωτού περάσουμε στην επόμενη φάση. Πρώτα απ' όλα θα λάβει τον λόγο η κυρία Μπέκενταμ, πρόεδρος της ΑΦΤΕΑ, που είναι Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενώσεων Γυναικών όσον αφορά την ε, ε, Αλία και η κυρία Μπέκενταμ που είναι επικεφαλής μιας οικογενειακής εκμετάλλευσης ε, η ίδια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα λάβει τον λόγο η κυρία Μπέκενταμ. Την καλωσορίζω βέβαια πρώτα. Dank u wel. Geachte leden van de commissie Visserijbeleid. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αλληλείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να πω δύο λόγια για την ακτέα που είναι το δίκτυο για τη, το οποίο εκπροσωπούμε, δίκτυο γυναικών. Είμαστε γνώμονες σε εσά για το γεγονός ότι μας προσφέρετε τη δυνατότητα να πούμε δύο λόγια για την ακτέα και για τα αποτελέσματα πως δίκτυο καταφέραμε να πετύχουμε μέχρι σήμερα. Η ΑΚΤΕΑ οφείλει την ύπαρξη της σε ένα πρόγραμμα ερευνητικό που ξεκίνησε από την Κάτια Φονγκούτ με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της διοργάνωσης διαφορετικών εκδηλώσεων, συνεδριάσεων σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες ερεύνησε η Κάτια για την κατάσταση των γυναικών όσον αφορά τις υδατοκαλλιέργειες. Δόθηκε παρότρινση σε πολλές γυναίκες να ακολουθήσουν τα θετικά βέλτιστα παραδείγματα και να μάθουν από άλλες. Το πιο σημαντικό ήταν όμως ότι έπρεπε να συνειδητοποιήσουν και συνειδητοποίησαν τη σημασία της ίδιας ε, της ε, δουλειάς τους, ε, της εργασίας τους. Και όταν κάνω λόγο για λύση εδώ, δεν κάνω λόγο μόνο για τον μικρό αριθμό γυναικών που ενεργά συμμετέχουν στις αλληλευτικές δραστηριότητες ή στην υδατοκαλλιέργεια, αν ενώ τις γυναίκες που ασχολούνται και με την πώληση των προϊόντων αλλά και με την ε, επισκευή, το μπάλωμα των δικτυών. Υπάρχουν και πολλές άλλες που πίσω από τα σκηνικά εργάζονται αθόρυβα και αόρατα όσον αφορά τις οικογένειές τους ε, έχουν και την ε, παρακολούθηση πληστηριασμών, ε, δημοπρατήσεων, τις επαφές με τράπεζες. Είναι η ραχοκοκαλιά όσον αφορά τις δραστηριότητες στο επίπεδο της στεριάς, τις στεριανές δραστηριότητες. Όταν λοιπόν ε, έληξε αυτή η περίοδος, η πρώτη περίοδος, αποφασίστηκε τις επαφές που είχαν ήδη ε, καλλιεργηθεί να τις ε, συνεχίσουν και να τις διευρύνουν ακόμα περισσότερο. Έτσι η ΑΚΤΕΑ ιδρύθηκε στην, στη συνέχεια στην Αγκώνα στην Ιταλία. Αποτελείται το δίκτυο από εθνικά, περιφερειακά, τοπικά δίκτυα γυναικών από 11 διαφορετικές χώρες. Η ΑΚΤΕΑ λοιπόν καταβάλει προσπάθειες για την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στην αλία και για την ίση μεταχείριση των γυναικών. Μέσω της υλοποίησης της οδηγίας 2010-41 από όλα τα κράτη-μέλη και του σεβασμού αυτής της οδηγίας. Αυτή η οδηγία προβλέπει την ίση μεταχείριση ανεξάρτητων γυναικών και ανδρών οι γυναίκες, οι Γαλλίδες γυναίκες έχουν το καθεστώς αυτό και είναι υπόδειγμα ήδη για τις υπόλοιπες γυναίκες. Μέχρι στιγμής ισχύει αυτό μόνο για τη Γαλλία. Για τις άλλες χώρες οι οδηγίες για τις εργαζόμενες ή συνεργαζόμενες γυναίκες ε, ε, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί πλήρως. Το νομικό καθεστώς δεν είναι επαρκές, ε, δεν επαρκεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα, ένα πρώτο βήμα το χρειάζονται οι γυναίκες για να συνεχίσουν να καταβάλουν τις προσπάθειές τους, θα δοθεί μεγαλύτερη κοινωνική προστασία και θα δοθεί και δυνατότητα να επεκταθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση. Παράλληλα καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες να συνεργάζονται σε οργανώσεις αλλιέων και στην λήψη αποφάσεων, στο επίπεδο λήψης αποφάσεων. Εδώ η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γυναικών αλλιέων από τις διαφορετικές χώρες και περιφέρειες είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Στην Αγκώνα το Προεδρείο συγκροτήθηκε και υπάρχει και μια ενημερωτική επιστολή αγγλικά και γαλλικά από την Ακτέα για τις δραστηριότητες του. Τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια τοπικών χορηγών υπήρξαν παρεμβάσεις δικές τους των ίδιων των γυναικών και αυτές ε, οι συνεδριάσεις, αυτά τα συνέδρια έχουν στο επίκεντρό τους ε, την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων. Ενθαρρύνονται, παρατρύνονται οι γυναίκες ε, να, διατηρηθούν, να διατηρήσουν την απασχόλησή τους ώστε να διατηρηθούν οι εκμεταλλεύσεις, οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και οι δραστηριότητες αυτές. Περνάμε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα οι γυναίκες είναι καταπληκτικές γεφυροποιοί για να γεφυρώσουν καταστάσεις και να μπορέσουν να επιβιώσουν οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ε, αποφασίζοντας υπέρ αηφόρων μεθόδων. Πολλές φορές ε, η αλληλεία δεν είναι το επαρκές μέσο για την ε, επιβίωση και διαβίωση. Χρειάζονται όμως περαιτέρω δραστηριότητες και το γνωρίζουν οι γυναίκες αυτό ε, οι δικές μας συνεδριάσεις είχαν θετικές επιπτώσεις ε, για την διασφάλιση και διατήρηση των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην παράκτια περιοχή. Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ των γυναικών αλλιέων οδήγησε στο ο αριθμός των γυναικείων οργανώσεων να αυξηθεί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία. Ακούμε μέσω των μηνυμάτων που φτάνουν στην ακτέα για την υλοποίηση αυτής της οδηγίας και έχουν, έχει ληφθεί απόφαση να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών να υλοποιήσουν αυτή την οδηγία που προανέφερα. Θα δώσω κάποια παραδείγματα για τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές ενεθάρρυναν τα μέλη της ΑΚΤΕΑ με το παράδειγμα των γυναικών που δημιούργησαν δίκτυο στη Γαλλικία το κατάφεραν να, να δημιουργήσουν ένα δίκτυο και να προσχωρήσουν ε, στην Περιφερειακή Ένωση. Παρότι οι Πορτογαλίδες γυναίκες ε, επιτελούν το ίδιο έργο, την ίδια εργασία, δεν έχουν ακόμα καταφέρει να αποκτήσουν αυτό το καθεστώς. Οι Γαλλικιανοί εφοπλιστές και πλειοκτήτες ε, έχουν, αντιμετωπίζουν και ένα θέμα παράνομης, απασχολούν παράνομα και εποχιακά αλλοδαφού εργαζόμενου. Αυτό είναι μια απειλή για τι ίδιε τι γαλλικιανέ γυναίκε. Στην Ολλανδία, από την οποία προέρχομαι, οι γυναίκε ε, αλληλεί, έχουν δημιουργήσει μια αγορά νοπού ψαριού. Το Σάββατο προσφέρονται αυτά τα προϊόντα, νοπά ψάρια, δείχνουν οι γυναίκες πώς καθαρίζονται τα ψάρια από τα λέφια και τα κόκαλα και πώς μπορούν να μαγειρευτούν με τον καλύτερο πιο νόστιμο τρόπο. Αυτή η αγορά συνεισέφερε σε εμά να ανοίξουν δρόμοι και ατραπή ώστε προϊόντα από την περιφερειακή αυτή αλληλεία να πολλούνται και να διοχετεύονται στην αγορά. Ήρθαν σε επαφή ε, και σε σχέση με τις Ολλανδές γυναίκες αλληλείς και από πλευρά και της Βόρειας Ιρλανδίας και με την Ακτέα υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις καθαρισμού ψαριών και μαγειρεύματο ψαριών και εκεί. Οι πρακτικές γνώσεις αυτών των γυναικών αλλιέων ήταν η καλύτερη διαφήμιση που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί για αυτά τα προϊόντα. Οι γυναίκες καλλιεργήτριες ε, οστρακοκαλλιεργιών στην Ορλεόν ε, αποφάσισαν να προσχωρήσουν και εκείνες σε τέτοιου είδου δράσεις. Μπορούσαν ε, οι καταναλωτές να δουν πώς ε, τρέφονται και πώς καλλιεργούνται αυτά τα οστρακόδερμα για να μπορούν μετά να συλλέγονται και να απολούνται στην αγορά. Είχαμε αυτές τις δραστηριότητες και σε συνεδριάσεις και εκδηλώσεις της ΑΚΤΕΑ και είδαμε ότι και από πλευρά της Ισπανίας με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε αυτές. Με αυτά νομίζω ότι δόθηκε ε, σε αδρές γραμμές ε, η εικόνα του τι γίνεται σήμερα σε σχέση με οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Υπάρχουν όμως πολλά προσκόμματα και εμπόδια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές γλώσσες στο ίδιο το δίκτυό μας και αυτό είναι ένα και δεν υπάρχει υποστήριξη από πλευράς των ανδρών, των οργανώσεων και συλλόγων των ανδρών αλλιέων ή από πλευράς ε, του κράτους. Το πιο σημαντικό είναι ότι έπρεπε να επιβιώσει η ακτέα χωρίς επιχορηγήσεις και κρατικές ενισχύσεις. Οφείλουμε πολλά σε επιστήμονες και ανεξάρτητους που μας βοήθησαν να τα καταφέρουμε με τόσο μικρά, τόσο μικρά κονδύλια που έχουμε να επιτελέσουμε το έργο μας. Τώρα όμως ήρθε η χρονική στιγμή να περάσουμε σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο και να ε, ασχοληθούμε κυριότερα με αυτά τα θέματα. Οι στρατηγικές για την ισότητα των γυναικών πρέπει να οδηγήσουν να ξεκινήσουν τέτοιου είδους δίκτυα, ώστε να βελτιωθεί ο ευδιάκριτος ρόλος των γυναικών, να γίνει πλέον ορατός και να είναι ευδιάκριτος και να μην είναι αόρατες οι γυναίκες. Είναι πεισμένη η ακτέα ότι ήρθε η χρονική στιγμή να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικών, γυναικείων οργανώσεων, ώστε να υπάρξει η διεύρυνση εθνικών, περιφερειακών, τοπικών δικτύων γυναικών, η διαδικτύωσή τους, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ανταλλαγή εμπειριών, να μπορέσουν να παρατηρηθούν οι γυναίκες να συνεισφέρουν όσον αφορά την αλία, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στους εαυτούς τους, να δουν ότι αξίζει τον κόσμο τρόπο να καταβάλουν αυτές τις προσπάθειες και είναι σημαντικό και για τον τομέα και να δούμε ποιες δυνατότητες θα υπάρχουν για την περαιτέρω επιμόρφωση και κατάρτιση για τις γυναίκες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες ότι η δουλειά τους για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις έχει μεγάλη σημασία για την ίδια την οικογενειακή εκμετάλλευση αλλά και για την διασφάλιση των δραστηριοτήτων στην αλληλεία συνολικά. Η ακτέα θέλει να διαδραματίσει ένα ρόλο σε αυτή την πιο επαγγελματική πλέον μορφή δράσης και να αποτελέσει μια πραγματικά επαγγελματική οργάνωση οι γυναίκες στην ίδια την αλληλεία δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν τίποτα αν πάρει αυτή την οργάνωση, τι πάρουν αυτή την οργάνωση άντρες ή γυναίκες που θα είναι εκτός συστάμενοι και δεν θα εμπλέκονται στα θέματα της αλληλεία, δεν θα γνωρίζουν τίποτα για την αλληλεία, δεν θέλουμε εκείνοι να μας αφομοιώσουν ή να μας εντό εισαγωγικών αποκτήσουν. Θέλουμε εμεί ε, αυθύπακτα να συνεχίσουμε να δρούμε. Και πίσω από κάθε εκμετάλλευση να ξέρουμε ότι βρίσκονται οι γυναίκε. Ευχαριστώ. A continuación, ε, tiene la... Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια για 8 λεπτά θα λάβει τον λόγο και σας παρακαλώ να τηρήσετε τα χρονικά όρια. Η κυρία Νατάδια είναι πρόεδρος ε, της Αγαμάδα, μιας ένωσης γυναικών που ασχολείται με, τις, με την συλλογή οστρακόδερμων το Δεκέμβριο 2007 ε, και είχαμε την, ε, το Forum of Fishing ε, Peoples και έτσι λοιπόν για 8 λεπτά σας δίνω τον λόγο και σας καλωσορίζω και εσάς κυρία Λαϊνέ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα ήθελα καταρχάς πριν ξεκινήσω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ σε αυτή την ακρόαση. Είμαι σίγουρη ότι θα προκύψουν ιδέες που θα αξιοποιήσουμε για να αναλύσουμε καλύτερα την κατάσταση και να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Ως πρεσιδέν, ως πρόεδρος της ε, Ένωσης της Γαλλικίας Οστρακός Συλλεκτριών θα ήθελα να μιλήσω για την ε, η συλλογή των οστράκων στη Γαλλικία είναι μια κοινότητα στην οποία ο τομέας αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η γυναίκα έχει ειδικό βάρος συγκριτικά με τους υπόλοιπους τομείς της αλίας. Αναμφισβήτητα η Γαλλικία έχει μια άρρηκτη σύνδεση με την θάλασσα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πάνω από 80 κοινότητες διαφόρων πληθυσμιακών μεγεθών έχουν πολύ στενές σχέσεις με τη θάλασσα. Ο αλληλευτικός κλάδος στη Γαλλικία αυτή τη στιγμή διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, συμβάλλει στη διατήρηση του πληθυσμού στην επικράτεια αυτή, ενώ αναπτύσσονται έτσι και άλλοι ε, τομείς. Το 10% του ΑΕΠ της Γαλλικίας ε, οφείλεται αποδίδεται σε αυτόν τον ε, αλλιευτικό τομέα. Κάτι το οποίο το έχει μόνο η Ισλανδία. Εάν μιλήσουμε για την καλλιέργεια οστράκων και τη συλλογή οστρακόδερμων γενικότερα, θα δούμε ότι έχει πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία στη δική μας κοινότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα και πιο πρόσφατα στοιχεία της κεντρικής διοίκησης, χάρη σε αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα φτάνουμε ε, σε ένα κύκλο εργασιών 75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίων, ετησίως για πάνω από 10.000 τόνους παραγωγής. Μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε ε, την ε, συλλογή οστράκων από τον αλλιευτικό στόλο αλλά και την ε, συλλογή οστράκων χειρονακτικά. Η πρώτη γίνεται μέσα από τη βάρκα, τον, τον, το αλλιευτικό σκάφος και είναι μια δραστηριότητα την οποία κάνουν κυρίως οι άνδρες. Η δεύτερη γίνεται ε, κυρίως από τις ε, γυναίκες. Έχουμε εισοδήματα για 5.000 ανθρώπους. Από αυτό ζουν 5.000 άνθρωποι στην Γαλλικία και το 90% αυτών των 5.000 ανθρώπων είναι γυναίκες. Ε, συλλέγονται λοιπόν τα όστρακα στις αμόδες ακτές χειρονακτικά, χωρίς κανένα στόλο είναι ουσιαστικά μια γυναικεία δουλειά στη Γαλλικία και οι οστρακοσυλλέκτριες ουσιαστικά είναι, σύμβολο διότι συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητάς μας. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς ε, λειτουργούν, τι ακριβώς κάνουν οι οστρακοσυλλέκτριες. Έχουν ενώσεις, οργανώσεις και ε, εκεί γίνεται η παραγωγή. Εκεί γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος των πόρων. Γίνεται σχεδιασμός της παραγωγικής διαδικασίας βάσει του σχεδίου εκμετάλλευσης που έχει προτείνει η κεντρική διοίκηση. Σε αυτό το σχέδιο περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις της ε, οικονομικής αυτής δραστηριότητας, από την αρχή μέχρι και τη συλλογή του προϊόντος. Έχουμε ε, το κιδόνι στις διάφορες ε, ποικιλίε. Μιλούμε για το ερυθρό, το λεπτό, το ιαπωνικό ή αυτό το οποίο στα ισπανικά ονομάζεται μπαμπόσα. Σήμερα στη Γαλλικία έχουμε 1134 αλλιευτικά ε, πάρκα ε, καλλιέργεια στις διάφορες περιοχές και στις διάφορες ζώνες. Σήμερα αυτό το επάγγελμα είναι αναγνωρισμένο. Εξού και υπάρχει νομοθεσία που ρυθμίζει τον κλάδο, ρυθμίζει τον επαγγελματικό χαρακτήρα αυτής της ε, δραστηριότητας είναι μέρος της ευρύτερης οικογένειας της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επομένως, πολύ συχνά πολλές οστρακοσυλλέκτριες είναι αυτές που ζουν την οικογένειά τους. Και βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η δραστηριότητα. Ουσιαστικά λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός της οικονομίας στην Γαλλικία. Ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν. Δώσαμε πάρα πολλούς αγώνες και πραγματικά συμμετείχαμε σε πάρα πολλές μάχες για να πιστοποιηθούν όλα αυτά και να γίνουν αποδεκτά από όλους. Οι οστρακοσυλέκτριες ε, εφήρμοσαν προγράμματα ανάπτυξης, οικονομικά προγράμματα και προγράμματα βελτίωσης της οργάνωσής τους. Χρειάστηκε να αλλάξουν την οτροπία τους η κάθε μία ξεχωριστά. Ε, πίστηκαν και πλέον είναι εκείνο τόπο ε, ότι είναι ε, ανάγκη να προχωρήσουν σε συλλογική δράση. Έχουν συλλογική νοοτροπία, ε, δεν ακούγονται πολλέ κατά τόπου φωνέ, αλλά μιλούν με μία φωνή για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Και γι' αυτό πέτυχαν στόχους από κοινού οι συλλογικότητέ τους, στόχου που δεν θα είχαν ποτέ καταφέρει η κάθε μία ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν να τα τονίσουμε όλο αυτό. Μιλούμε δηλαδή για ε, δράσεις σε ενώσεις, για εργασιακές ε, ε, ενώσεις και επαγγελματικές ενώσεις. Έχουμε τις συντεχνίες των αλλιέων. Αυτά είναι όργανα που βοηθούν τις οστρακοσυλέκτριες να κάνουν μια πιο συστηματική δουλειά και να αξιοποιήσουν καλύτερα τους πόρους. Καλό θα είναι επίσης να μιλήσουμε για την δημιουργία ενώσεων και οργανώσεων σε ε, κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Η δική μας οργάνωση, η Αγκαμάρ, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εμείς θέλουμε να είμαστε η φωνή που θα εκφράσει τις ανάγκες του κλάδου. Να ζητήσουμε τα να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά μας και να απαιτήσουμε τη βελτίωση ε, της δραστηριότητας αυτής. Η Αγκαμάρ ουσιαστικά ε, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καταρτίζει, υπάρχει και κατάρτιση και μεταφέρει στην κεντρική διοίκηση όλα τα αιτήματα, τα παράπονα αλλά και τις ανάγκες ε, των οστρακοσυλλεκτριών στη Γαλλικία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία η σημερινή για να τονίσουμε και το εξής. Οι οστρακοσυλλέκτριες ελέγχουν αυτή τη διαδικασία από την εξόριξη του οστράκου μέχρι και την ε, θέση του προς πώληση. Πολύ συχνά μεγάλο μέρος του κέρδους όμως παραμένει στα χέρια των διανομέων και όσων ε, θέτουν σε εμπορία τα προϊόντα. Καλό θα είναι να έχουμε περισσότερους ελέγχους στην ανιχνευσιμότητα του προϊόντος, ώστε επιτέλους οι οστρακοσυλέκτριες να έχουν τη σωστή αμοιβή που τους αξίζει, διότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Από εκεί και πέρα ε, ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η κατάρτιση όλου αυτού του τομέα, του κλάδου. Ως Αγκαμάρ, ως Ένωση, οργανώνουμε μαθήματα για να, για να έχουμε καλύτερη κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα. Ε, κάνουμε λοιπόν τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Πέρα από την κατάρτιση Κάτι που θα πρέπει να καλύψουμε επίσης είναι το θέμα της πρόληψης των κινδύνων. Να σας επισημάνω το εξής. Στη χειρονακτική αυτή συλλογή οστράκων, η μεθοδολογία, τα εργαλεία είναι ε, θα τα χαρακτηρίζω σχεδόν πρωτόγωνα, δηλαδή δεν επηρεάζουν καθόλου ε, το περιβάλλον, δεν το επηρεάζουν καθόλου αρνητικά. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το ότι δηλαδή δεν λειτουργούν σε βάρος του περιβάλλοντος. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι χρειάζεται κανείς να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες για να χειριστεί αυτά τα ελευτικά εργαλεία ε, τα οποία ε, υπάρχουν και έτσι πολύ συχνά υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Ε, πέρα από αυτό, εάν σε αυτό προσθέσουμε τις επικίνδυνες μετεωρολογικές συνθήκες, τα πολύ εξαντλητικά ωράρια, βλέπουμε ότι οι συνέπειες στην υγεία των οστρακοσυλλεκτριών είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε ε, παθήσεις ε, του μυοσκελετικού συστήματος και επαγγελματικά νοσήματα. Και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στον τομέα της πρόληψης όλων αυτών των κινδύνων. Γι' αυτό και ως Αγκαμάρ έχουμε σχεδιάσει και έχουμε φτιάξει δύο συγκεκριμένες στολές για τις ηλέκτριες, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν, να δουλέψουν καλύτερα, αλλά να είναι και καλύτερα προστατευμένες. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για την ε, πρόληψη ε, κινδύνων. Τώρα, επανερχόμενοι σε αυτό το θέμα της ε, συλλογικής δράσης και της δημιουργίας ενώσεων, θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι είναι καλό να ανταλλάξουμε εμπειρίε και να ε, αποκοινούν να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας και τη βελτίωση των ε, εργασιακών ε, συνθήκων. Η Αγαμάρ λοιπόν είναι μέλος του Παγκόσμιου Φόρου, Φόρουμ των ανθρώπων που ασχολούνται με την αλληλία, που είναι μια διεθνής οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν διάφορε ενώσει μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Έτσι μαθαίνουμε τι γίνεται σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας σε αυτό το φόρουμ ε, διότι ε, βρίσκουμε σημεία στήριξης για να προχωρήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση του κλάδου μας. Ως Ένωση λοιπόν, ως οργάνωση θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και είναι και πολύ σημαντικό το σχέδιο νόμου ε, για την βιώσιμη αλληλεία θα πρέπει η κοινή αλλιευτική πολιτική να λάβει υπόψη της πόσο σημαντική είναι η ερασιτεχνική αλληλεία, αν θέλετε, και τα ωφέλη της ε, για τη διατήρηση των διαφόρων οικοσυστημάτων, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ε, βιοτόπων. Αυτού του είδους η αλληλεία συμβάλλει ε, και στην οικονομική δραστηριότητα. Έτσι ο κλάδος μπορεί να επιβιώσει. Άρα χρειάζονται μέτρα, ένα πακέτο μέτρων που να λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Η αναγνώριση των ενισχύσεων για όλο αυτό το θέμα ε, είναι πολύ καλή. Ουσιαστικά αποτελεί στήριξη για εμάς. Η χειρονακτική συλλογή οστράκων αυτή τη στιγμή έχει δεν μπορεί να πει κανεί ότι έχει μείνει στο απειρόβλητο. Βεβαίω και έχει επηρεαστεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Έχουμε πολύ μεγάλη μείωση των πωλήσεων. Έχουμε χαμηλέ τιμέ επίση στην αγορά. Η κατάσταση λοιπόν είναι αρκετά ε, δυσχερείς και δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον του κλάδου. Ωστόσο θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να μαχόμαστε, να απαιτούμε τα δικαιώματα ε, τα οποία χρειάστηκαν τόσα πολλά χρόνια ε, για να κατοχυρώσουμε. Θα ενώσουμε τις φωνές μας ζητώντας τη βελτίωση των μελλοντικών προοπτικών για τις εργαζόμενες στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λαϊνό. Στη συνέχεια και παρακαλώ να σέβεστε τον το όριο του χρόνου. Όταν θα έχετε ε, ολοκληρώσει το όριο του χρόνου θα χτυπάμε το σφυράκι και θα πρέπει να τερματίζετε. Η κυρία Καρίς Κάνια στη συνέχεια, πρόεδρος ε, της ε, Ουμάρ Αζόρες, μια ένωση για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών της ε, Ένωσης ε, Αλίας ε, των Αζωρών, Ίσων Αζωρών στην Πορτογαλία. Και όσον αφορά το ΡΑΚΑ των δυτικών παράκτιων περιοχών, έχετε τον λόγο παρακαλώ κυρία Κάνια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή είναι μια ευκαιρία <clears throat> όπου στοχεύουμε να διατυπώσουμε κάποια ερωτήματα για την ιδέα για την βιοτεχνική αλληλεία που κοινωνικά και οικονομικά έχει ιδιαίτερο βάρος και σημασία. Και η πολυμορφία των δραστηριοτήτων των γυναικών στη βιοτεχνική αλληλεία αποτελεί πραγματικά μια δουλειά ένα, μια εργασία που είναι αόρατη, άφαντη από τη μια πλευρά και έχει και ένα, μια συνιστόσα αορατών δραστηριοτήτων από την άλλη. Και θα πρέπει να, ε, να γνωρίσουμε την αξία της εργασίας των γυναικών στην Αλία και μέσω της ε, ε, ενωσιακής δραστηριότητας σε συλλόγους και ενώσεις να μπορέσει αυτό να διαχυθεί και να γίνει γνωστό στην Ευρώπη. Η βιοτεχνική αλία έχει μια κοινωνική και οικονομική σημασία ιδιαίτερη στις διαφορετικές χώρες χώρες ε, της Ευρώπης ε, και στις ε, νησιωτικές περιοχές όπως τις Αζόρες. Αποτελεί έναν ε, τομέα που πέρα από τη διασφάλιση της ποιότητας ε, των ψαριών, των αλλιευμάτων για την ανθρώπινη κατανάλωση, συνεπάγεται και πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Όταν κάνουμε λόγο για τη βιοτεχνική αλληλεία, κάνουμε λόγο για τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται. Για την αλληλεία μιλάμε για γυναίκες και άνδρες. Κάνοντας λόγο για την βιοτεχνική αλληλεία μιλάμε για τον ρόλο των γυναικών γυναικών που έχουν πριτανεύοντα ρόλο εκεί. Οι γυναίκες όσον αφορά τη βιοτεχνική αυτή ε, αλληλεία, μέρος αυτής της εργασίας ε, είναι ορατό και άλλο μέρος ε, δεν είναι ορατό και δεν το γνωρίζουμε αποτελούν ένα πολυάριθμο, μια πολυάριθμη ομάδα οι γυναίκες σε αυτή την δραστηριότητα, στη βιοτεχνική αλία, με ρόλους και δραστηριότητες που συνδέονται με τη ζωή της αλίας στις κοινότητες, τις παράκτιες και τις νησιωτικές. Αυτή η πραγματικότητα τονίζεται και αφορά διαφορετικούς ρόλους και δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι γυναίκες στη βιοτεχνική αλληλεία. Τα τελευταία χρόνια μέσω της ε, αναβάθμισης και αξιολόγησης ε, των γυναικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε μέσω από τις δράσεις που αναπτύχθηκαν από θεσμικά όργανα, ε, ομάδες, ενώσεις, συλλόγους, δίκτυα γυναικών στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένων και χωρών και περιοχών νησιωτικών όπως είναι οι Αζόρες. Σε αυτή τη διαδικασία έχει καθοριστική σημασία η εμφάνιση οργανώσεων γυναικών στην Αλία, όπως η περίπτωση της ΑΚΤΕΑ, Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναικών στην Αλία, που ανέπτυξε ε, εργασία, δουλειά σε αυτό το πεδίο, συνενώνοντας διαφορετικές ενώσεις ε, και συλλόγους, όπως ε, και από διαφορετικές χώρες, όπως και την Πορτογαλία. Τα τελευταία χρόνια πρέπει να τονιστεί ο ρόλος στο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και στην Άμπα, στην ε, νήσο Τερσέρα των Αζωρών, στην Ήλιας ε, Ενρέτζη, τα νησιά στο δίκτυο Ένωση Γυναικών της Αλίας στις Αζόρες και την Ουμάρ Αζόρες. Στην Πορτογαλία, στι Αζόρε και στη Μαδέρα η βιοτεχνική αλληλεία έχει πολύ μεγάλο κοινωνικό βάρο ε, και οι γυναίκε έχουν τονίσει τον ρόλο του μέσω προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αναβάθμιση, αξιολόγηση, αναγνώριση τη δουλειά του ε, και ενδυνάμωση του ρόλου του. Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, το να συμμερίζονται τις εμπειρίες τους ε, και τα προβλήματά τους οι γυναίκες ε, μέσα στους διαφορετικούς περιφερειακούς χώρους και τομείς, ε, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και προκλήσεις, αποτελεί μια βάση για να οικοδομήσουμε μια πορεία προς την προάσπιση της βιοτεχνικής αλίας, συμπεριλαμβάνοντας γυναίκες και άνδρες σε αυτόν τον σημαντικό κοινωνικό-οικονομικό τομέα στην Ευρώπη. Θεωρείται επίσης σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος και η σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην Αλία σε όργανα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, όπως είναι ε, τα συμβουλευτικά αλλιευτικά συμβούλια, περιφερειακά ε, ε, συμβούλια για την αλληλεία, καθώς επίσης και να τονίσουμε επίσης και τη σημασία της ανταλλαγής και ε, εμπειριών και απόψεων μεταξύ των ενώσεων γυναικών ε, στην Αλληλεία στην Ευρώπη. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις ε, και σκέψεις. Πρώτον, είναι σημαντικό να προαγάγουμε την παρουσία και τη συμμετοχή των γυναικών στα θεσμικά όργανα, στη, λήψη αποφάσεων, στις οργανώσεις και οργανισμούς των επαγγελματιών της Αλίας. Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη και η σημασία να διασφαλίσουμε ένα χώρο και αναγκαία υποστήριξη για να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες των λήψεων αποφάσεων στο πολιτικό επίπεδο. Δεν επαρκεί να σκεφτούμε στη σημασία της συμμετοχής των γυναικών είναι επίση αναγκαίο ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε όρου και προποθέσει ώστε αυτή η συμμετοχή να μπορεί να πάρει σάρκα και οστά και να ε, γίνει πραγματικότητα. Τρίτον, είναι αναγκαίο να προαγάγουμε, να προωθήσουμε την ανταλλαγή μέσων και προγραμμάτων και σχεδίων για να διασφαλίσουμε την ε, ε, κατάρτιση και εκπαίδευση των γυναικών, επενδύοντας ε, στην αυτοεκτίμησή τους, στην αναβάθμισή τους, στο να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο και τη σπουδαιότητα που έχει η δουλειά τους. Να γνωρίζουμε, τέλος, το θέμα του να γνωρίζουμε τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την αλληλεία και τομεακά και τον ε, που πρέπει να ταυτίζονται ανάλογα με το φύλλο, ξεχωριστά για τις γυναίκες. Να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται αυτό και θα συλλέγονται αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Και η ανάγκη να επικαιροποιηθεί η έρευνα να, είναι, να εξυγχρονιστεί η έρευνα για τις ε, δραστηριότητες των γυναικών στην Αλία και να υπάρξουν μελέτες που θα συνταχθούν. Και για την ενημέρωση από πλευρά ΑΚΤΕΑ έχει συνταχθεί ε, ε, αντίστοιχη μελέτη και φαίνεται ότι υπάρχει ανάγκη σήμερα να γίνει μια μελέτη που θα δίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο χωρών, κρατών μελών και σε επίπεδο περιφερειών την εικόνα, την πραγματική εικόνα της συμμετοχής και εργασίας των γυναικών στην Αλία σε κάθε μια από τις χώρες μας και περιφέρειές μας και στην Ευρώπη συνολικά, σαν μια μορφή να διασφαλίσουμε την καλή ε, προαγωγή του προγραμματισμού των μέτρων και σχεδιασμού των μέτρων, ώστε να αναβαθμιστεί η βιοτεχνική αλία και η συμπερίληψη των γυναικών παράλληλα με τους άνδρες σε αυτόν τον τομέα πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ. Muchas gracias eh, a eh. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ γιατί δεν ξεπεράσατε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λέσλι Ντάδη, εκπρόσωπο του δικτύου γυναικών της Βορείου Θάλασσας. Η καταγωγή της είναι από το Φράζεμπουργκ, στη βορειοανατολική Σκοτία είναι μέλος της οργάνωσης αυτής εδώ και τρία χρόνια. Και θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα για την εμπειρία που έχει αποκομίσει από τη συμμετοχή της ε, στην Ένωση αυτή και από τις συζητήσεις ε, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων και πιο συγκεκριμένα για το Περιφερειακό Γνωμικό, Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Βορείου Θάλασσας. δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο 2003 ως αποτέλεσμα ε, προγράμματος ε, για τις ε, κοινότητες της Βορείου Θαλάσσης να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που θα δώσει μια ενωμένη φωνή στις ε, γυναίκες και ένα μέσο για εξέβριση λύσεων σε κοινά προβλήματα. Έχουμε περίπου 60 μέλη στα κράτη της Βορείου Θάλασσας ε, και επικοινωνούμε ηλεκτρονικά και ε, με διασκέψεις. Βεβαίως μπορεί να γίνει μέλος όποιος ενδιαφέρεται από την αλλιευτική κοινότητα για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής και εργασίας και να αναπτυχθούν δυνατότητες επιχειρήσεων και κατάρτισης. Είμαστε μέλος ε, της οργάνωσης ΑΚΤΕΑ που δίνει στις ε, γυναίκες ε, δυνατότητες δικτύωσης σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθούμε ε, βασικά να εξασφαλίσουμε ότι οι συνέπειες οι κοινωνικές και οι οικονομικές της αλλαγής της αντιευτικής πολιτικής, ποσοστώσεις ε, και τάκ μέγιστο προβλεπόμενο αλλίωμα ε, να ακούγεται η φωνή μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο και Επίσης αυτό γίνεται με, μέλη στα ΡΑΚ, στα συμβούλια, τα περιφερικά, τα γνωμοδοτικά. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά θέματα λαμβάνονται υπόψη και κάθε ομάδα εργασίας να τα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα αυτά. Επίσης έχουμε προσελκύσει κονδύλια από το Ηνωμένο Βασίλειο και για να γίνει μια μελέτη σχετικά με την αλία. Ε, στο δικό μας ε, το Συμβούλιο Εργαζόμαστε για να αναπτύξουμε δεσμούς με την Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης για παροχή στοιχείων, εκθέσεων και εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ελευτική πολιτική και να εξεταστούν παράγοντες που θα συμβάλλουν στην αξιοπιστία της αλίας και να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αλλαγές στην αλία. Βεβαίως, έχουμε ένα κοινό πρόβλημα που είναι η χρηματοδότηση υποστήριξη όπως έχουν όλα τα δίκτυα γυναικών. Ε, βρήκαμε όμως υποστήριξη οικονομική για να μπορέσουμε να προσχωρήσουμε στο Πελαγικό Συμβούλιο. Ως, ε, ως μητέρα ε, και σύζυγος αλλιέων πελαγικών με χρόνο τώρα στα χέρια μου θέλω να ασχεληθώ πολύ περισσότερο για το μέλλον του κλάδους. Επίσης, έχω εντυπωσιαστεί από τις συλλογικέ γνώσεις και κατανόηση για να προετοιμαστούν συστάσεις για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αποθέματα τα πελαγικά αντιμετωπίζονται από προγράμματα μακροπρόθεσμα διαχείρισης. Πρέπει να δούμε πώς θα επανασχεστούν αυτά τα προγράμματα ούτως ώστε να έχουν καλύτερη απόδοση ως προς τα ε, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες για τον κλάδο. Αυτό σημαίνει μεγιστοποίηση των αλλιευμάτων όταν αυτό καθίσταται βιώσιμα δυνατό. Θα πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να συμμετέχουν στην εργασία των περιφερειακών συμβουλίων. Μπορώ να συμμετέχω σε συζητήσεις δεν, δεν αγωνιζόμαστε μόνο για την ζωή μας. Είναι ένας τρόπος ζωής, υπήρξε για γενναίες και ελπίζω για πολλές επόμενες γενναίες. Αλλά πολλοί λέει νέοι στρέφονται προς τη θάλασσα λόγω της αβεβαιότητας των ποσοστώσεων ως γυναίκες ε, μπορούμε επίσης ε, να κάνουμε τις ευρύτερε κοινότητες να συμμετέχουν στη συζήτηση και θα πρέπει επίσης να δούμε και τις ε, διάφορες βιομηχανίες που υπάρχουν στον τομέα, διότι πάρα πολλές θέσεις εργασίας παραδοσιακές χάθηκαν. Αυτό ήταν καταστροφικό. Ε, βεβαίως δεν απασχολούνται τόσο πολύ στη θάλασσα διότι ε, περιλαμβάνονται στον κλάδο μηχανικοί συγκολητές, ε, ναυπηγοί, αυτοί που η παραγωγή δικτύων, αυτοί που βάφουν τα πλοία κλπ. Το προϊόν απαιτεί πάρα πολύ ποιότητα. Το προϊόν χρειάζεται φωνή και θα πρέπει οι γυναίκες να έχουν τέτοια φωνή και να εξασφαλίσουμε οι συνέπειες οικονομικές των περικοπών των ποσοστώσεων να λαμβάνονται υπόψη στις τελικές αποφάσεις. Θα πρέπει τα περιφερειακά συμβούλια ε, να συνεργάζονται μαζί με τις ομάδες εργασίας και την Εκτελεστική Επιτροπή, να μοιράζονται τις ιδέες μεταξύ των κρατών μελών. Η συμβολή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προωθηθεί όλος ο κλάδος. Αλλά τι γίνεται όταν ψηφίζονται οι συστάσεις. Πάρα πολλές συστάσεις απορρίπτονται διότι δεν εξετάζονται εντελεχώς, ε, διότι ε, ε, οι εκθέσεις οι εκθέσεις επιστημονικές έρχονται σε σύγκρουση με τις συστάσεις μας. Πάρτε πάντως χάρη τις πρόσφατες συζητήσεις για την Ρέγκα στην Βόρειο Θάλασσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μήπως μπορείτε να μιλάτε ε, κάπως πιο αργά, λέει η Πρόεδρος, γιατί διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα. Συνεχίστε παρακαλώ. Άρατε παραδείγματο χάρη τις πρόφασες συζητήσεις για τη ρέγγα της Βορείου Θάλασσας λόγω αναθεώρησης από την ΆΙΣΕΣ σχετικά με το επίπεδο αναπαραγωγής φαίνεται ότι τα ΤΑΚ μέγιστη προβλεπόμενο αλίευμα για το 2009 και 2010 είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ε, η ICS βρήκε το σφάλμα που είχε κάνει στην αρχή ε, του έτους ε, και έχουν αναθεωρηθεί για το 2010 τα ΤΑΚ προς τα πάνω κατά 19%. Ε, υπήρξε ε, μια, ε, ένα 4% μείωση το 2010 και περαιτέρω αύξηση 15% θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στις αναθεωρημένα στοιχεία. Αλλά δυστυχώς οι συστάσεις του Συμβουλίου του Περιφερειακού του Πελαγικού απορρίφθηκαν. Ε, καμιά φορά η συμβολή μας, η συνεισφορά μας αγνοείται. Ελπίζω ότι αντιπροσωπεύοντας ε, τις αλλιευτικές κοινότητες στο Περιφερειακό, Περιφερειακό Συμβούλιο ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ε, διαφορά, ότι θα μπορούμε να διαμορφώσουμε κάτι για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντριάννα Σελεστίνη, πρόεδρο της Ένωσης Γυναικών Πινελόπη, ε, γυναίκες της Αλίας της ε, περιοχής της Αγκώνα στην Ιταλία. Θα μας μιλήσει για το Μεσογειακό Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Βλέπετε, βλέπετε κυρία Επίτροπε ότι έχουμε πολλούς εκπροσώπους από ε, διάφορα περιφερειακά συμβούλια. Είναι αντιπρόεδρος της ΑΚΤΕΑ αλλά και πρόεδρος της Επιτροπής για την Ισότητα των Ευκαιριών στην περιοχή της. Έχετε το λόγο παραλαβώ. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε εδώ την ε, ένωσή μας ε, και την, να μιλήσουμε για την κατάσταση των γυναικών ε, που εκπροσωπούνται σε αυτήν. Όλοι κάνουν λόγο για αυτόν τον τομέα που είναι πολύ παραγωγικός και ξέρουμε όμως ότι βρίσκεται στα χέρια των ανδρών. Παρ' όλα αυτά οι γυναίκες εκπροσωπούνται πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα, παρότι και με, με μη πολύ ευδιάκριτο τρόπο. Ε, ως συνεργάτριες ε, σε αυτές τις επιχειρήσεις τις οποίες ε, εργάζονται ή στην Αλία. Φαίνεται μόνο άνδρες να εργάζονται. Αυτό είναι ο ευδιάκριτος χαρακτήρας των δραστηριοτήτων τους. Όμως και οι γυναίκες ε, που ε, κάνουν τόσες πολλές δουλειές διαδραματίζουν και εκείνες ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Αλία. Εμείς στην Ιταλία έχουμε την εμπορευματοποίηση, την ε, διάθεση στο εμπόριο, έχουμε υπόψη και αναλαμβάνουμε τα διάφορα γραφειοκρατικά, τα διάφορα γραφειοκρατικά καθήκοντα πρέπει να μπορέσω να ολοκληρώσω. Είναι αδύνατον όμως με αυτή την ταχύτητα να συνεχίσετε. Λυπούμε. Και οι διερμηνείς ε, θα πάθουν νευρική κρίση αν ε, συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και πρέπει να διασφαλίσω και την υγεία των διερμηνέων. Θα σας δώσω δύο λεπτά παραπάνω αλλά να μιλάτε λίγο πιο αργά παρακαλώ. Εντάξει, τότε λοιπόν θα μπορέσω να έχω δύο λεπτά περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, έλεγα ότι οι επιχειρήσεις ε, στον τομέα της ε, αλληλείας ε, και της δραστηριότητας Λοιπόν, να δω αν θα το καταφέρω με αυτή την ταχύτητα. Οι γυναίκες έχουν τα καθήκοντα εμπορίας των αλλιευμάτων, τα τη γραφειοκρατία, ε, τα θέματα των συνεταιρισμών και των δικτύων και επειδή οι άνδρες λείπουν, βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα κατά τη διάρκεια όλων των ημερών, εργάσιμων ημερών της εβδομάδας και έτσι οι γυναίκες ε, αναλαμβάνουν τις υπόλοιπες δουλειές ε, και βλέπουμε ότι σε σχέση με τις ακτές τις παράκτης περιοχές οι ίδιοι οι πλειοκτήτες είναι κυβερνήτες, είναι καπετάνιοι στα σκάφη τους και οι γυναίκες στην πλειοψηφία τους εργάζονται σε συνεταιρισμούς ε, ε, όπως και έχουν και τους πιο διαφορετικούς ρόλους. Δεν έχουν όμως ένα νομικό καθεστώς που να τις προστατεύει οι γυναίκες. Και για αυτές τις γυναίκες που συνεργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις ε, είναι ανάγκη να υπάρξει αυτό το καθεστώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως νοικοκυρές, σαν γυναίκες που εργάζονται στο σπίτι τους και δεν έχουν κάποιο άλλου είδους δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είναι πεισμένες ότι ε, επιπλέον ασκούν κάποιες ε, περισσότερες δραστηριότητες πέρα από αυτές ε, που ασκούν ως ε, νοικοκυρές. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό το πλαίσιο πραγμάτων. Ξεκινά η δουλειά τους όταν ε, δένουν τα πλοία το πρωί και όταν φτάνουν τα αλλιεύματα και ξεφορτώνονται, ξεφορτώνονται και μετά περνάνε ε, κάνουν χιλιόμετρα από το λιμάνι για να μπορέσουν να πολιθούν στις καλύτερες τιμές και μετά γυρίζουν στα νοικοκυριά τους, στα σπίτια τους και επομίζονται όλες τις άλλες δραστηριότητες. Βλέπετε ότι οι πολυσχηδείς, οι πολύμορφες εργασίες που επομίζουν οι γυναίκες είναι πάρα πολλές και πολύ κουραστικές. Πρέπει να αναγνωριστεί η ποιότητα και το είδος και η αξία αυτής της εργασίας. Έτσι οι γυναίκες θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν και να θεωρήσουν γνωρίζουν με διαφορετικό τρόπο τη δουλειά τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Θα γνωρίζουν καλύτερα τις ευθύνες ε, που επομίζονται και στον τομέα που συμμετέχουν και εργάζονται. Βελτίωση και στο κοινωνικό πλαίσιο. Λείπει ο χρόνος όμως πολλές φορές ε, και πολλές φορές ε, δεν γνωρίζουν ποια είναι η αξία αυτής της δουλειάς και βλέπουμε ότι οι γυναίκες εργάζονται σε αυτόν τον τομέα με αυτόν τον τρόπο. Ιδιαίτερα όμως οι γυναίκες στην Αγκώνα αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σύλλογο, αυτή την ένωση, να γίνει γνωστό το έργο τους και να το αναγνωρίσουν όλοι. Δημιουργήθηκε λοιπόν η Ένωση Πινελόπη, ο Σύλλογος Πινελόπη Γυναίκες στην Αλία. Στόχος είναι να αναγνωριστεί ο κοινωνικός ρόλος και η δραστηριότητα των γυναικών στις δικές μας παράκτιες περιοχές, αναζητώντας διασφακα... να κατοχυρώσουν και να εγγυηθούν ε, οι δραστηριότητές τους για να, γνωρισ... να αναγνωριστεί η αξία στον τομέα αυτό της εργασίας τους και να μην ε, απολεστεί η παράδοση και να μπορέσουμε να να μάθουμε από αυτήν. Είναι ευθύνη λοιπόν που επομίζονται οι γυναίκες όλα αυτά μέχρι να καταλήξουμε και στην ίδια την ε, οικογενειακή εκμετάλλευση ή επιχείρηση που πρέπει να εξοπλίζεται και με, πληροφορική, με τον εξοπλισμό για την πληροφορική και να έχει σχέσεις και με άλλες ε, επιχειρήσεις και δίκτυα να μπορέσει να αναπτυχθεί ε, στο η γυναίκα και ως άτομο αλλά και ως μέλος μιας κοινωνίας. Πράγματι η Πινελόπη, Πενέλοπη βρίσκεται και εκείνη ως μέλος της ακτέα και από πλευράς των γυναικών στην Αλία συμμετέχουμε σε αυτό το πλαίσιο. Όλες οι γυναίκες λοιπόν που είναι στην ακτέα από όλες αυτές από την Κύπρο, από την Ιταλία, βλέπουμε ότι δεν έχουμε ένα νομικό καθεστώς. Οι άλλες γυναίκες στην ακτέα έχουν ένα νομικό καθεστώς. Θεωρούνται συνεργάτριες των αλλιευτικών αυτών μονάδων στις οποίες εργάζονται. Δεν βρισκόμαστε εμείς λοιπόν σε ίσο επίπεδο με τους άνδρες, ενώ εργαζόμαστε στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό ε, σοβαρή έλλειψη. Επίσης, σε σχέση με τη συμμετοχή σε μία εκμετάλλευση ε, με πλήρη ε, χαρακτηριστικά, υπάρχει διαφορά μεταξύ γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλλιευτικών εκμεταλλεύσεων. Σε μία γεωργική εκμετάλλευση η συμβία, η σύζυγος ή η βοηθός ε, του άντρα που είναι επικεφαλής μπορεί να αναγνωριστούν με ένα νομικό καθεστώς, να αναγνωριστεί το νομικό τους καθεστώς, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο στην αλλή. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο λοιπόν ανδροκρατίας θα έλεγα, ακραία υπερβολικής ανδροκρατίας εις βάρος των γυναικών. Θα πρέπει να βγουν από την σύραγγα της άτυπης εργασίας, μη αναγνωρισμένης εργασίας οι γυναίκες και να αποκτήσουν το καθεστώς ε, της, ε, των εξειδικευμένων εργατριών. Ε, δεν υπάρχει ούτε και χρόνος αρκετός που να απομένει στις ίδιες τις γυναίκες από πλευράς ελεύθερου χρόνου. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσει αυτή η πραγματικότητα να αλλάξει. Πολλές γυναίκες από την Καλαβρία και την Σικελία δημιουργούν παρόμοια δίκτυα όπως το δικό μας της Πινελόπης. Έχουμε διαφορετικές ενώσεις λοιπόν και συλλόγους στην περιοχή μας. Διασφαλίζονται λοιπόν τα δικαιώματα των γυναικών εκεί όπου υπάρχουν ενώσεις και σύλλογοι. Χρειαζόμαστε όμως και υποστήριξη για να μπορέσει να γνωστοποιηθεί αυτό το έργο, να υπάρξει συλλογή πληροφοριών, να υπάρχει μεγαλύτερο θα έλεγα ε, περισσότερο περισσότερο αλληλέγγυο πνεύμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την ε, δραστηριότητά μας ε, ε, να συνδεόμαστε με δίκτυα και να δημιουργούμε ενώσεις. Διαφορετικά η νοοτροπία δεν θα αλλάξει και η πραγματικότητα δεν θα αλλάξει. Πρέπει οι γυναίκες να αναγνωριστούν και να αναγνωριστεί ο ρόλος και η σημασία τους μέσα από τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι εύκολη η δουλειά αυτή. Είναι σημαντική σημαντικό το έργο της ενωσή μας, αλλά αντιμετωπίζουμε μια ολόκληρη σειρά προσκομμάτων και εμποδίων θεσμικά, διότι αποτελείται ο τομέας αλληλεία όχι μόνο από τους άνδρες και ε, εργαζόμενους άνδρες αλληλεί, αλλά επίσης έχουμε και την οικονομική κρίση και την νομοθεσία που ευνουχίζει και οδηγεί σε αδιέξοδο πολλές προσπάθειες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν παραδόσεις ε, που είναι διαφορετικές όσον αφορά την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη υποστήριξη και προαγωγή αυτών των θεμάτων. Επικεντρωνόμενοι τώρα στα, στο Συμβούλιο ε, στο, για τη Μεσόγειο, το, η συνιστόσα του ε, φίλου θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη σε αυτό το συμβουλευτικό όργανο. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες ώστε να μπορέσουν να αναγεννηθούν, να δημιουργηθούν περισσότερες οργανώσεις και ενώσεις όπως ε, η Πινελόπη. Και με το θέμα αυτό της αναγνώρισης το ίδιο πρέπει να πούμε ισχύει και για τις γυναίκες που ζουν στην απέναντι όχθη της Μεσογείου, στη βόρεια ακτή δηλαδή της Αφρικής. Και ολοκληρώνω πρόεδρε λέγοντας ότι οι γυναίκες στον τομέα της Αλίας από τη Γαλλία λένε ότι όταν μια γυναίκα παντρεύεται, δεν παντρεύεται μόνο έναν άντρα, αλλά παντρεύεται ένα ολόκληρο τομέα και τις παραδόσεις του. Και γι' αυτό πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον χαρακτήρα και τη δραστηριότητα των γυναικών που εργάζονται σε αυτό το τομέα και να τις εισακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Κάτια Φραγκούδη, η οποία δεν είναι εδώ, ε, τότε θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Μονίκ Φιλίπ. Α, από ό,τι μου ενημερώνουν επίσης δεν ε, μπορεί να είναι μαζί μας γιατί ε, ε, ένα σκάφος από το λιμάνι από το οποίο προέρχεται έχει εξαφανιστεί και υπάρχουν δύο αγνοούμενοι και πρέπει να σταθεί δίπλα στις ε, των δύο αγνοούμενων. Λοιπόν, η κυρία Φραγκούδη αντικαθιστά την κυρία Μονίκ Φιλίπ ε, και είναι ερευνήτρια σε θέματα κοινωνικά στο Πανεπιστήμιο της Μπρέστ. Καλημέρα σας εξ ονόματος της Ομοσπονδίας της γαλλικής ε, των γυναικών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημόσια κρόαση και για την πρόσκληση που απίφθινε σε αυτήν ε, την Ομοσπονδία. Εφόσον η Μονίκ Φιλίπ δεν είναι εδώ παρούσα, θα διαβάσω την παρουσίασή της. Θα προσπαθήσω να μην ε, μιλάω γρήγορα. Ίσως το επιτύχω, γιατί δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά η γλώσσα εργασίας, μας, εργασίας μου. Η ε, Γαλλία, οι γυναίκες αυτού του περιβάλλοντος έχουν από το 1960 ε, δημιουργήσει μια ένωση ε, και αργότερα στη δεκαετία του 90 για να μοιραστούν την εμπειρία τους, να ε, επιτύχουν την εξέλιξη του σε επαγγελματική τους θέσης και να μπορέσουν να καταλάβουν στην οικογένεια και στην επιχειρήση τη θέση που τους ανήκει λόγω της εργασίας τους. Ε, πρόκειται για γυναίκες αλλιέων, αλλά όχι για ε, γυναίκες αλληλείς οι οποίες εκπροσωπούνται από συνδικάτο. Οι γυναίκες αυτές ε, λοιπόν ε, στάνθηκαν αυτήν την αναγκαιότητα για να ανταλλάξουν απόψεις, για να συναντώνται και για να ακουστεί η φωνή τους. Έχουμε ως μέλη στην Ομοσπονδία Γυναικών και Οικογενειών Ναυτικών ε, η Association Charentaise από τη Βρετάνη μέχρι τη χώρα των Βάσκων, ε, ε, μια ένωση στην Μεσόγειο, μια στην Κορσική και μια στην Λεκάνη του Τό. Ε, η δημιουργία του 1998 για το καθεστώς ε, του συζύγου ή της συζύγου ε, συνεργάτριας και εδώ η Γαλλία είναι πρωτοπόρος. Αυτή η θέση, αυτό το καθεστώς έδωσε μια όθηση στην οργάνωση των γυναικών. Αρχικά, οι γυναίκες που επέλεξαν αυτό το καθεστώς δεν ήταν πολυπληθείς διότι δεν ήταν κάτι το υποχρεωτικό. Αλλά από το 2008 το καθεστώς αυτό ε, του συζύγου, του συμβίου, του συνεργάτη είναι υποχρεωτική για κάθε ε, σύζυγο ή ε, συμβία που συμβάλλει στην αλλιευτική επιχείρηση και όλο και περισσότερες γυναίκες υπάρχουν. Έχουμε τώρα περίπου 900 γυναίκες που έχουν επιλέξει το καθεστώς αυτό. Το καθεστώς αυτό για την οστρακοκαλλιέργεια ε, και την αλία ε, δίνει δικαίωμα για ατομική σύνταξη των γυναικών, αλλά ανοίγει ε, και τις πόρτες των επαγγελματικών οργάνων όταν ο σύζυγος δεν θέλει να παρουσιαστεί. Μερικές γυναίκες βρίσκονται επικεφαλής των οργανώσεων ανδρών. Επίσης το καθεστώς είναι δικαίωμα σε επαγγελματική κατάρτιση που χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Κατάρτισης για την Αλία. Στο τέλος του 2007 το πιστοποιητικό του συζύγου, της συζύγου συνεργάτη ε, της βιοτεχνικής επιχείρησης έχει δημιουργηθεί. Είναι ένα δίπλωμα εθνικό που βοηθάει ε, της Συνδίας να επιτελέσουν καλύτερα την εργασία τους στην αλλιευτική επιχείρηση. Το κόστος της κατάρτισης αναλαμβάνεται από επαγγελματικού οργανισμούς ενώ οι γυναίκες των ναυτικών δεν μπορούν να ωφεληθούν από αυτή την χρηματοδότηση και πρέπει να βρούνε άλλοι μόνο οι ε, συνεργάτες ε, σύζυγοι. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένες από αυτές τις ε, πρόοδους για αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, η συλλογική εργασία της οργάνωσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν ε, έχουν αναγνωρισμένη θέση ούτε οι ενώσει, οι οργανώσει, ούτε οι ομοσπονδίε. Τα μέσα είναι ανεπαρκή για να μην μπούμε ανύπαρκτα, για να μπορέσει ε, μια ομοσπονδία να λειτουργεί καλά και να επικοινωνεί με τρόπο αποτελεσματικό με τα μέλη του δεκτύου ε, και με όλα τα άλλα όργανα αφετέρου. Η έδρα ε, είναι στο, στην κατοικία της Προέδρου του Σώματος Αλίας και αυτό ισχύει για όλες ε, τις ε, ενώσεις ακόμα και την ακτέα. Τα μέσα, τα υλικά είναι περιορισμένα και η ατομική συνδρομή οικονομική των μελών απαιτείται συχνά. Οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες αλλά είναι χρειάζονται έξοδα και αυτό αποκλείει τις γυναίκες που είναι από άπορες οικογένειες. Χρειάζονται λοιπόν ειδικά και μόνιμα χρηματοδοτικά μέσα. Τα έξοδα των δράσεων που προτείνεται, η εκπόνηση των σχεδίων, η κατάρτιση των στελεχών, η οργάνωση σε σεμινέρια, η επικοινωνία, η συμμετοχή σε διάφορα όργανα και οργάνωση ενός μιας μόνιμης ομοσπονδιακής ε, μονάδας ε, έχουν εκτιμηθεί και παρουσιαστεί στις εθνικές αρχές που αρνήθηκαν αυτή τη χρηματοδότηση. Για να κατανοήσετε καλύτερα τις δυσκολίες μας, θα σας δώσω ένα πραγματικό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ε, της Ένωσης ε, των Γυναικών ε, του Μπασάνταρ Κασό, από όπου προέρχεται εκεί η Μονίκ Φιλίπ, που παρουσιάστηκε για χρηματοδότηση στον άξονα 4 του Αλληλευτικού Ευρωπαϊκού Ταμείου. Στο πλαίσιο λοιπόν της, του τοπικού προγράμματος, η Ένωση θέλει να δημιουργήσει μια συλλογική συνεργατική εταιρεία ε, για την δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες που έρχονται από το θαλάσσιο περιβάλλον ε, και ε, για άτομα με ειδικέ ανάγκες και για αναβάθμιση των προϊόντων που αλλιεύονται στον Μπασάνταρ Κασό με συνταγές για το μαγείρεμά τους και την ε, δημιουργία βιβλίων, συνταγών, επικοινωνία με σχολές κλπ. Το πρόγραμμα που προτάθηκε φαίνεται πολύ σημαντικό στις, στα όργανα λήψεως αποφάσεων που μας συμβούλευσαν να την πραγματοποίηση μιας τεχνικο-οικονομικής μελέτης που θα έπρεπε να αναλάβει η οργάνωσή μας και να την χρηματοδοτήσει που θα κοστίσει 50.000 ευρώ ε, ποσό που δεν ε, διαθέτει ε, η οργάνωσή μας, διότι αν την είχαμε δεν θα χρειαζόμασταν τη βοήθεια του Ταμείου. Ή στο μέτρο που η οργάνωση δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή τη μελέτη, να αρχίσουμε εκπονώντας ένα βιβλίο συνταγών και να δημιουργήσουμε εργαστήρια για το μαγείρεμα των προϊόντων της θάλασσας ε, με θελοντικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση ο άξονας 4 του Ελιευτικού Ταμείου του Ευρωπαϊκού θα μπορούσε να δώσει μια βοήθεια, μια ενίσχυση. Κλείνοντας, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν εξαιρετικές ιδέες για την αναβάθμιση των αλληλευτικών προϊόντων, για την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν την δυσκολία αναγνώρισης της συλλογική συνεργατική τους εργασία ε, και αντιμετωπίζουν την έλλειψη των χρηματοδοτικών μέσων. Και θα πρέπει συνεχώς να δικαιολογούν την εργασία που έχει γίνει, ε, που συχνά κρίνεται ως μη αξιόπιστη από τα περισσότερα όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να δώσω το λόγο στην κυρία Νόρα Πάρκε, συντονίστρια της Οργάνωσης Παραγωγών της Ιρλανδίας, της Οργάνωσης Αλλιέων του Κίλιμπεξ. Η κυρία Πάρκε εργάζεται στην οργάνωση αυτή από το 2005 και ασχολείται κυρίως με τη διαχείριση της θέσης σε εμπορία του καβουριού και την ενημέρωση των μελών ως προς τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση των συνθηκών αγοράς. Η Ένωση αυτή συνεργάζεται στενά με άλλες οργανώσεις, τοπικές, εθνικές αλλά και διεθνείς. Κυρία Πάρκε, έχετε το λόγο για 8 λεπτά περίπου. Γεια σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας απευθύνω το λόγο σήμερα σε αυτήν εδώ την ακρόαση. Με εξέπληξαν πάρα πολλές παρουσιάσεις ε, ε, που, έκαν, οι προηγούμενες ομιλήτριε. βλέπω ότι έχετε πολύ μεγάλο δυναμισμό. Είστε γυναίκες ε, πάρα πολύ δραστήριες στον τομέα τη αλίας και σα συγχαίρω γι' αυτό. Εγώ είμαι υπάλληλο στην οργάνωση αλίου του Κίλιμπεκ και είμαι συντονίστρια σε θέματα καβουριού. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση αλλιέων παραγωγών στην Ιρλανδία και ασχολούμαστε κυρίως με το πελαγικό, το βίνθο πελαγικό αλλά και το ε, καφετί, το καστανό καβούρι. Εγώ είμαι βιολόγος και ε, ουσιαστικά όλη μου τη ζωή την έχω περάσει ε, ασχολούμενη με τα θέματα αυτά αφού η οικογενειακή επιχείρηση των γονιών μου είχε να κάνει επίσης ε, με τα όστρακα και τις ε, ε, καλλιέργειες αυτές. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια συγκεκριμένη περίπτωση που δείχνει ότι ε, μπορούν οι γυναίκες να είναι πολύ αποτελεσματικές. Είχαμε ένα πολύ τεράστιο πρόβλημα, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια λόγω της κακής διαχείρισης αυτού του είδους της αλλιευτικής δραστηριότητας. Ξέρετε, την αλία του καβουριού την κάνει η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βορειοδυτική ε, Γαλλία. Δηλαδή, τρία διαφορετικά δικαιοδοτικά όργανα επισέρχονται εκεί και έχουμε και ε, μια συνιστόσα εγχώρια αλλά και εξωχώρια. Και σε κάθε ένα από αυτά τα όργανα και δημιουργούνται πολλές περιπλοκές. Ανοιχτή πρόσβαση λοιπόν, επομένως τεράστια αύξηση της αλλιευτικής δραστηριότητας, της αλλιευτικής δυνατότητας τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2007, 2008 και μετά. Γι' αυτό έχουμε αυτό που παρατηρείται από το 2007 και μετά είναι μια κατακόρυφη πτώση ε, της ζήτησης άρα και των τιμών. Άνθρωποι από διαφορετικές χώρες αλλιεύουν λοιπόν αυτό το είδος καβουριού και επικοινωνούν ελάχιστα μεταξύ τους και γι' αυτό έχουν όλοι μπει σε αυτό το παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών ο ένας στον άλλον. Οι συμμετέχοντες ε, στις οργανώσεις στην ε, κάστοτε χώρα κατηγορούν ε, τους ομολόγους τους ε, στην άλλη χώρα. Έλλειψη επικοινωνίας, επομένως έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτά ήταν τα στοιχεία που χαρακτήριζαν την κατάσταση. Έχουμε το ελάχιστο μέγεθος εκφορτώσεων και έχουμε και τα σκάφη 15 μέτρων. Όλες αυτές είναι προϋποθέσεις, αλλά δεν επαρκούν για τον έλεγχο αυτής της πολύ σημαντικής αλλιευτικής δραστηριότητας ε, γνωρίζαμε την απουσία επικοινωνίας και προσωπικά ως συντονίστρια για θέματα του καβουριού στην Ιρλανδία, ήρθε σε επαφή επανειλημμένως με τους αλληλείς στις άλλες χώρες και πιο συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και γι' αυτό ξεκαθαρίστηκε στο μυαλό μου η ανάγκη ε, να καθίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν για τα προβλήματα που έχουν γιατί είναι κοινά σε όλους τα προβλήματα αυτά. Επομένως, με συναδέλφους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία ε, οργανώσαμε μια σύσκεψη τον Ιανουάριο του 2010 την πρώτη φορά. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά αυτή ε, τον Ιανουάριο του 2010 όπου συναντήθηκαν οι πιο μεγάλοι παράγοντες, οι πιο σημαντικοί φορείς και αντάλλαξαν απόψεις. Ε, η σύσκεψη αυτή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ξεπέρασε κατά πολύ τουλάχιστον τις δικές μου προσδοκίες προέκυψαν ε, δύο πολύ σημαντικές προτάσεις από την ε, συνάντηση αυτή. Πρώτον, οι αλληλείς να μειώσουν τις εκφορτώσεις κατά 25% ε, και στη συνέχεια να έχουμε μια διεθνική προαγωγή θέση σε εμπορία και μάρκετινγκ. Γιατί ξέρετε, τελικά στην Ευρώπη δεν καταναλώνεται πολύ καβούρι και αν αυξηθεί η ζήτηση τότε θα έχουμε ε, πολύ θετικά αποτελέσματα, πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Ε, έγιναν περαιτέρω συσκέψεις στο Παρίσι, στο Εδιμβούργο, για να ε, μεταφερθούν οι προτάσεις αυτές στον ευρύτερο κλάδο, υψηλή συμμετοχή σε αυτές τις συναντήσεις παρατηρήθηκε. Επίσης, ε, με αυξημένο επίπεδο συνένεσης. Και το Μάρτιο συναντηθήκαμε για άλλη μια φορά στο Παρίσι και οριστικοποιήσαμε τις λεπτομέρειες όσων είχαν συζητηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης σύσκεψης αλλά και ε, τη συνάντηση στο Εδιμβούργο. Είχαμε εκπροσώπους από την Ουαλία, τη Σκοτία, την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, από την ε, ακτή της Βορείου Αγγλίας, από το, ε, από το Isle of Man και από διάφορες άλλες περιοχές. Οι προσπάθειες που έγιναν για τη μείωση των εκφορτώσεων κατά 25% μιλούν από μόνες τους. Βλέπετε στη διαφάνεια τις ε, τιμές, η κόκκινη γραμμή για το 2009 ε, και βλέπετε τη σημαντική αύξηση της τιμής για το 2010. Παρόλο που δεν το τήρησαν όλοι αυτό, ε, έγινε. Είχαμε σημαντική μείωση και αυτό δείχνει ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η πρόταση αυτή, η οποία δούλεψε τελικά. Και φάνηκαν και τα αποτελέσματα. Βεβαίως η τιμή δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα. Οι ίδιες οι χώρες επιτάχυναν τις προσπάθειές τους, εξέτασαν τις στρατηγικές διαχείρισης που ακολουθούν και σίγουρα θα υποβάλουν καλύτερα ε, σχέδια διαχείρισης για τα επόμενα έτη. Τώρα, τι μπορώ να πω για το μέλλον. Τρία πράγματα. Τρία έψιλον ε, αν θέλετε. Επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία, να λαμβάνει χώρο επικοινωνία σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και ε, θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετάσχουν σε αυτήν και να την ενθαρρύνουν ε, ε, γκρινιάζοντας συνεχώς και παρενοχλώντας με την κλασική αυτή τεχνική ώστε να έχουμε περισσότερο, ε, περισσότερη επικοινωνία μεταξύ μας. Νομίζω ότι αυτή η συνεργατική προσέγγιση είναι προς όφελος όλων. Όλοι κερδίζουν από αυτήν. Για πρώτη φορά συνειδητοποίησαν οι παριστιάμενοι ότι όλοι αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση και δεν τα πηγαίνει καλύτερα η μία χώρα συγκριτικά με την άλλη. Όλοι πλήττονταν και όλοι θα είχαν πολλά ωφέλη να αποκομίσουν ε, μιλώντας με τους συναδέλφους τους, με τους ομολόγους τους και υιοθετώντα κοινή δράση. Αυτή τη στιγμή η δραστηριότητα αυτή, δηλαδή η προσπάθεια μείωσης των εκφορτώσεων, επηρέασε σημαντικά τον κλάδο, βοήθησε πολύ τη βιωσιμότητα, είχε λιγότερο αντίκτυπο στα αποθέματα. Άλλωστε, με τη μείωση των εκφορτώσεων, τα, ο στόλο περνά λιγότερο χρόνο στη θάλασσα, άρα χρειάζεται λιγότερο καύσιμο, λιγότερα δολώματα, ε, λιγότερο αντίκτυπο στο βαθύβιο και βυνθοπελαγικό ε, περιβάλλον. Και έτσι επιτυχάνονται και καλύτερε τιμέ. Το βασικό μήνυμα λοιπόν είναι να καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι, να μιλήσουμε για τα προβλήματά μα και να δούμε τι δράση μπορούμε από κοινού να πάρουμε πριν αναγκαστούμε να προχωρήσουμε προχωρήσουμε σε ρύθμιση νομοθετική. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πάκε. Στη συνέχεια θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και μια συζήτηση στην οποία προφανώς όλοι μπορείτε να συμμετάσχετε. Από πλευρά των Ευρωβουλευτών ζήτησε τον λόγο ο Ρωμέβα πρώτος. Παρακαλώ κύριε Ρωμέβα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για όλες τις ε, παρεμβάσεις, εισηγήσει. Ήταν πολύ εμπλουτιστικές και σίγουρα θα πρέπει να πω ότι ε, ήταν ε, σίγουρα επαρκέστατες. Θέλω να πω ότι αξίζουν την αναγνώρισή μας όπως η Γαλλικιανή Ένωση Βιοτεχνικής Αλίας. Είναι αναγκαίο να εκφράζονται τέτοιοι προβληματισμοί αλλά και εδώ να δούμε τα θέματα τα οποία τίθενται. Ε, μία απλή ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω στις διάφορες συναδέλφους εκπροσώπους των οργανώσεων. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε ευκαιρία να επισκεφθούμε μεταξύ άλλων και την περιοχή της χώρας των Βάσκων, όπου συνήθαμε με διαφορετικές διάφορες οργανώσεις γυναικών και εκεί διαπιστώνεται ένα πρόβλημα που επαναλαμβάνεται ως πρόβλημα σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ο αόρατος χαρακτήρας, ο μη ορατός χαρακτήρας της εργασίας των γυναικών στην αλληλεία άφαντος. Στην πρακτική όμως και το πιο ε, ανησυχητικό είναι αυτό, στη νομική πραγματικότητα ανύπαρκτος ρόλος των γυναικών, προστασία των γυναικών και όσον αφορά τις ε, άδειες, ε, τις απουσίες, την αποχώρηση από την εργασία. Είναι ακατανόητο ότι τόσες χιλιάδες άτομα, τόσες χιλιάδες γυναίκες που συνεχίζουν να εργάζονται και είναι θεμελιώδους σημασίας για τον τομέα της αλίας και για το έργο τα, τις ανάγκες της αλίας να είναι αόρατες και να εξακολουθούν να είναι απούσες. Ερώτηση λοιπόν, σε ποιο μέτρο και βαθμό εργάζεστε ή μπορεί να υπάρξει εργασία για να αντιμετωπιστεί αυτός ο αόρατος χαρακτήρας. Υπό το πρίσμα των ενώσεων και συλλόγων είναι κάτι πάρα πολύ αναγκαίο. Αλλά υπό το πρίσμα το νομικό και το νομοθετικό Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, για την κοινωνική ασφάλιση και αναγνώριση τη υπηρεσία εργασία, αυτέ οι κατηγορίε συμβάσεων που θα μπορούσαν πολλέ φορέ να δώσουν απαντήσει σε πολλέ από αυτέ τι δραστηριότητε είναι αόρατε, είναι ανύπαρκτε δυνατότητε. και σε πολλά άλλα μέρη τη Ευρώπη. Είναι κάτι γενικευμένο για τι γυναίκε αυτό. Και εν τέλει θα έπρεπε το νωρίτερο δυνατό να βρεθεί λύση για αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σάντσες Πεσέδο παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα ο ίδιος να συγχαρώ να συγχαρώ όλες τις εισηγήτριες που παρενέβησαν με ένα τόσο πολυσχηδές διαφορετικές απόψεις που είχαμε, πολυσχηδείς απόψεις και διαφορετικές τοποθετήσεις είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε τώρα η χρονική στιγμή που έχουμε και μια γυναίκα επίτροπο που είναι ε, γυναίκα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίτροπος, να υπάρξει δράση. Υπάρχει συνειδητοποίηση από πλευρά τη ε, και θέλω σε σχέση με αυτή την ε, πρωτοβουλία να συγχαρώ για την ανάληψή της. ο προβληματισμός μου είναι ο εξής θα αναφερθώ σε αυτά τα θέματα και σε σχέση με την Ένωση της Γαλλικίας, που είναι η κοινότητα που γνωρίζω περισσότερο. Εκεί η εξόριξη των οστρακοδέρμων είναι ε, ε, δραστηριότητα χιλιάδων ατόμων, πάρα πολύ έντονου χαρακτήρα όσον αφορά την εργασία και όσον αφορά τις πληροφορίες που έχω, η παραγωγή οστρακοδέρμων είναι επικεντρωμένη σε πολύ μικρή περιφέρεια, πολύ μικρή γεωγραφική επικράτεια. Μεγάλη προσπάθεια έρευνας θα πρέπει να γίνει για να μπορέσει να αυξηθεί και η παραγωγικότητα στο υπόλοιπο της Γαλλικίας. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να αυξηθεί αυτή η παραγωγικότητά παραγωγικότητά τους, δίνοντας μεγαλύτερα κίνητρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις δραστηριότητες και υποστήριξη. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση των γυναικών που εργάζονται στην οστρακοκαλλιέργεια και εξορρυκτική δραστηριότητα. Όσον αφορά την ανταλλαγή γενεών, την ανανέωση με νέες ε, ε, γυναίκες θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αναγκαίες προσαρμογές ε, για να υπάρξει εισαγωγή νέων γυναικών στην εργασία αυτή όσο είναι δυνατόν. Και τρίτον, αυτή η δραστηριότητα που αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και με τα υδατοκαλ... τις υδατοκαλλιέργειες και τα θαλάσσια πάρκα συνδέεται πολύ με τις περιβαλλοντικές ε, ε, ε, με περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέσεις. Τι γίνεται σε σχέση με τις δραστηριότητες σας αυτές μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πώς μπορούν να ενισχυθούν. Ευχαριστώ κυρία Μπιλμπάου παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω εγώ ίδια όλες τις ενώσεις και εκπροσώπους των ενώσεων αυτών που μας μίλησαν για τις διαφορετικές εμπειρίες και που μας ε, ανέφεραν και τα σχετικά με τα δίκτυά τους, όπως οι εκπρόσωποι από τη Γαλλικία για τον ορατό χαρακτήρα, ευδιάκριτο χαρακτήρα. Αυτή η συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι μία μικρή απότηση φόρου τιμή στι τόσε χιλιάδε γυναικών που εργάστηκαν ώστε να είναι δυνατόν στον κόσμο τη θάλασσα και η διασφάλιση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ίσω ε, επειδή ήταν μέρο και τη ίδια τη ζωή μου να ευχαριστήσω για αυτή τη συνεισφορά, για τη δημιουργία αυτών των δικτύων, για να αξιολογηθεί και να αναβαθμιστεί η δουλειά των γυναικών που εργάζονται και εργάστηκαν στις διαφορετικές μας χώρες, εργαζόμενες στη θάλασσα. Θέλω να υπενθυμίσω ένα πράγμα, επειδή εδώ έγινε λόγος για αυτή τη δουλειά που κάνουν στα λιμάνια οι γυναίκες, με τις διαφορετικές πραγματικότητες. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτές οι γυναίκες ε, πάντα εργάζονται και στα σπίτια τους, στον οικοκυριό τους, ως οικοκυρές αυτός ο αόρατος χαρακτήρας λοιπόν είναι διπλός αυτής της δουλειάς τους, μέσα στον οικοκυριό και έξω από τον οικοκυριό τους και χωρίς οποιαδήποτε αναγνώριση κιόλας για όλο αυτό το έργο που επιτελούν. Είναι σημαντικό τα βήματα τα οποία γίνονται, στα βήματα αυτά που κάνουμε να ληφθούν υπόψη αυτές οι πολυσχηδείς διαφορές στην πραγματικότητα, αλλά και ένα πράγμα που είναι σημαντικό, το βήμα που έγινε, ώστε οι γυναίκες σε σχέση με τη θάλασσα η εργασία τους να μην είναι βοηθητική, αλλά να είναι δουλειά αυτοτελής, μέσα από την οποία να μπορούν να ζουν με μισθούς αξιοπρεπείς αυτές οι γυναίκες. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να δημιουργηθούν πλήρη μεροκάματα για αυτές τις γυναίκες, να ξεπεράσουμε αυτή την έννοια που ακούσαμε του αόρατου, του μη ορατού και αναγνωρισμένου ε, έργου που δεν είναι βοηθητικό το έργο της γυναίκας αλλά είναι αυτοτελές και αυτούσιο. Ερώτηση λοιπόν, η Επίτροπος Δαμανάκη, υπό το πρίσμα ε, το δικό μου με σημαντικές συνεισφορές, θα ήθελα να ρωτήσω ε, για τις ενώσεις. Γνωρίζουν επαρκώς όλες ε, τις δυνατότητες ενίσχυσης τις, των οποίων μπορούν να τύχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν έχουν κάποια δυσκολία να στραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχυθούν για να βελτιωθεί η ζωή τους και η κατάστασή τους να βελτιωθούν τα πράγματα μέσω αυτών των διεργασιών, μέσα από αυτή τη συνεργασία και υποστήριξη της συνδρομής αυτής, της οποίες θα τύχουν. Δεύτερον, αν βλέπουν και αναγνωρίζουν ότι μέσα στη μεταρρύθμιση, αναρρύ, ε, μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής υπάρχουν δυνατότητες για να συνεισφέρουν ή να υπάρξει μια παρέμβαση ή πώς νομίζουν ότι μπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο για να μπορέσουν οι παρεμβάσεις αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές όσο αφορά την κοινή αλλιευτική πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάτια Φραγκούδη έχει ζητήσει το λόγο δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας, λέει η Πρόεδρος, και μετά η Νατάλια Λάινο. Η Κάτια πρώτα έχει το λόγο, παρακαλώ. όσον αφορά την αναγνώριση της εργασίας των γυναικών και κυρίως αυτήν την αόρατη εργασία σε επίπεδο κοινοτικό υπάρχουν ορισμένες οδηγίες που επιτρέπουν ακριβώς τα κράτη-μέλη αν θέλουν να τις μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο να αναγνωρίσουν την εργασία ε, του συζύγου ή της συζύγου συνεργάτιδας, ε, όπως έκανε η Γαλλία. Η ε, σύζυγος που συνοδεύει τον σύζυγό της είτε στην επιχείρηση την αλλιευτική είτε των οστρακοειδών. Και... Αλλά βεβαίω η κάθε χώρα αλλα βεβαιως η καθε χωρα εχει τα δικά της ασφαλιστικά ταμεία ως προς τον τομέα της Αλλία και δυστυχώς δεν διαθέτουμε καμία συνολική γενική μελέτη όσον αφορά στον κοινωνικό τομέα της αλίας γενικά. Αυτή τη στιγμή ε, δεν ξέρουμε για τους άνδρες, είναι δύσκολο να γίνει αυτό για τις γυναίκες. Αλλά όσον αφορά στην Ισπανία νομίζω ότι είναι πιθανόν η μόνη, το μόνο κράτος ε, που αναγνωρίζει, που παρέχει κοινωνική ασφάλιση στις γυναίκες, στην οικογένεια, στην ε, σύζυγο ή στα παιδιά που εργάζονται για την αλλιευτική επιχείρηση. Ε, στα άλλα κράτη η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και η Ισπανία έχει η ειδική κοινωνική ασφάλιση για την Αλία, όπως την Γαλλία, την Ελλάδα ή την Πορτογαλία, αλλά άλλες χώρες δεν έχουν. Δεν έχουμε μια τέτοια μελέτη γενική συνολική. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε τις οδηγίες της ευρωπαϊκές ε, στα εθνικά δίκαια. Όσον αφορά λοιπόν ε, στο γεγονός αυτό, οι γυναίκες είναι αόρατες, αλλά μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο, στην πρόκληση και να προωθήσουν τα δικαιώματά τους. Και όλες οι οργανώσεις των γυναικών εδώ δείξουν ότι δεν περίμεναν ούτε τις κρατικές ενισχύσεις, ούτε μια βοήθεια από κάποιον για να ιδρύσουν τις οργανώσεις τους, τις ίδρυσαν μόνες τους για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, διότι έχουν δικαιώματα και γενικά δεν το είπαμε εδώ, σε πάρα πολλές χώρες είναι χάρη στην κρίση της αλίας που οι γυναίκες ίδρυσαν τις οργανώσεις τους. Ήταν απόρρια της κρίσης στον τομέα της αλίας. Για να έρθω στην ερώτηση που έθεσε η κυρία εδώ μπροστά. Είναι αληθές ότι εργάζονται κατοίκον και εργάζονται και για την επιχείρηση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για ορισμένες γυναίκες ε, οι οποίες κάνουν πάρα πολλή δουλειά στο σπίτι τους ε, και στην επιχείρηση λογιστικά, τηλεφωνούν στον πελάτη. Είναι δύσκολο για αυτές να τα συμφιλιώσουν όλα. Είναι δύσκολο να πετήσουν μια αναγνώριση. Αλλά η διαδικασία όσον αφορά τις ενισχύσεις που δίνονται στις οργανώσεις των γυναικών δεν υπάρχει. Για την Ακτέα που είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο Ε, βλέπετε την κατάσταση. Οι τοπικές οργανώσεις μπορούν να επιτύχουν τοπικές ενισχύσεις, αλλά όταν πρόκειται για οργανώσεις εθνικές ε, δεν υπάρχουν. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, η οδηγία είναι σαφής στον άξονα 3, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τα δίκτυα των γυναικών. Αλλά αν τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να υποστηρίξουν τις οργανώσεις γυναικών όπως είναι η κατάσταση, κανείς δεν μπορεί να τις υποχρεώσει. Η Επίτροπη δεν μπορεί να τις έχουμε λοιπόν την, ε, την θέση, το καθεστώς του συζύγου ή της συζύγου. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση μεταφοράς της οδηγίας ε, και έχουμε, αλλά το κανονισ, τον κανονισμό σχετικά με τον Ταμείο Αλίας δεν μπορεί η, η, η Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη να αναγνωρίσουν ε, τις οργανώσεις των γυναικών αν έχουν εξοδεύσει τα ε, χρήματα αλλού. Μας μένει λοιπόν ο άξονας 4 του Ταμείου Αλίας, αλλά αυτά είναι για ειδικά προγράμματα, ειδικέ δράσεις που θα έχουν παρουσιάσει οι γυναίκες. Δεν είναι για υποστήριξη προς τις οργανώσεις αυτές καθεαυτές. Ίσως τώρα θα μπορούμε να σκεφτούμε πώς το επόμενο, ε, ο επόμενος κανονισμός, αν υπάρξει, θα μπορεί να λάβει υπόψη αυτό, δηλαδή να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι για τις γυναίκες. Αλλά σταματάει εκεί το πράγμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κυρία ε, Ναταλία Λάινο, παρακαλώ. Καλησπέρα και πάλι. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που μου θέσατε. Αναρωτηθήκατε αν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με την οστρακοκαλλιέργεια στη Γαλλικία. Όντως, η αυτόνομη κυβέρνηση της αυτόνομης κοινότητας της Γαλλικίας έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τη διαχείριση ε, της αλληλευτικής δραστηριότητας στη Γαλλικία. Αυτό είναι σαφές. Ωστόσο, να σας, πω, ε, να σας μιλήσω για ένα νούμερο. Είμαστε στο 10% της παραγωγής που έχουμε στις αμμώδεις ε, ακτές της Γαλλικίας. Δηλαδή, μπορούν όντως να υλοποιηθούν προγράμματα ευρωπαϊκά για να φτάσουμε στο 100% της αξιοποίησης των περιοχών αυτών. Από εκεί και πέρα τίθεται και το πρόβλημα της ηλικίας, της γύρανσης ε, του γυναικείου πληθυσμού, ο οποίος κατά μέσα όρο είναι 55 έως 60 ετών. Ο γυναικείος πληθυσμός που ασχολείται με αυτή την οστρακοσύλλογη και οστρακοκαλλιέργεια αν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε κάποια προγράμματα για να φτάσουμε στο 100% της παραγωγής, τότε νέες γυναίκες θα έμπαιναν σε αυτό το κλάδο και θα έβλεπαν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται. Θα ήταν κάτι το αποδοτικό από οικονομικής σκοπιάς για αυτές. Είναι σημαντικό βεβαίως να πούμε ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να συμφιλειωθεί με την οικογενειακή ζωή, γιατί το ωράριο είναι τετράωρο καθημερινά. Επομένως, εύκολα μια γυναίκα μπορεί μετά να ε, ασχοληθεί με την οικογενειακή της ε, ε, ζωή. Από εκεί και πέρα, έχουμε τις ζώνες C στην Γαλλικία. Έτσι τις ονομάζουμε, στην Φερόνα ή στην Παγιόν. εκεί δεν έχει γίνει πλήρης βιολογικός ε, καθαρισμός. Υπάρχει υπερφόρτωση ε, στο δυναμικό των παράκτιων περιοχών και ασκείται πίεση για να ε, χτιστούν, να κατασκευαστούν σωστές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων ώστε όλες οι επιχειρήσεις να έχουν δικές τους εσωτερικές μονάδες και να έχουμε σωστή παρακολούθηση της κατάστασης και να μην κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει. Από εκεί και πέρα, έχουμε κάποια πάρκα υδατοκαλλιέργειας. Αυτά υπάρχουν σε ατομική βάση, προσωπική βάση. Έχουμε τέτοια πάρκα στην ζώνη του Καρίλ, κατά κύριο λόγο και εκεί η έλεγχη είναι πιο άμεση. Ε, επειδή αυτό είναι ιδιοκτησία ιδιωτική, ε, την προσέχει καλύτερο ο ιδιοκτήτης της. Ενώ όταν κάτι είναι δημόσιο αγαθό, κοινό, ε, πολύ συχνά ο καθένας από εμά το παραγνωρίζει, δεν το προσέχει, δεν το φροντίζει τόσο πολύ. Εάν μια έκταση σου ανήκει σε ένα προσωπικά, τη φροντίζει την καλλιεργεί την κάνεις να αποδίδει 100% την προσέχει, την προστατεύει περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια μορφή πιο ε, σωστή, είτε μέσω συντεχνιών, είτε μέσω συνεταιρισμών. Δεν ξέρω, αλλά ε, να κάνουμε κάτι ώστε οι αμμώδεις ακτές όπου καλλιεργούνται και συλλέγονται αυτά τα όστρακα να φτάσουν στο 100% της δυναμικότητάς τους, της παραγωγής τους, όπως ήδη συμβαίνει με τα πάρκα υδατοκαλλιέργειας στο Καρίλ, τα οποία είναι ιδιωτικά, ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους και γι' αυτό εκεί έχουμε υψηλή αποδοτικότητα. 62 είναι περίπου οι συντεχνίες και συνεταιρισμοί στη Γαλλικία, με δεκάδες χιλιάδες γυναίκες, που ε, συμμετέχουν σε αυτούς τους συνεταιρισμούς συλλογής και καλλιέργειας οστράκων, πέραν των ανδρών που ασχολούνται με την αλλιευτική δραστηριότητα στην ανοιχτή θάλασσα με τον αλλιευτικό στόλο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πολλά και βεβαίως ζητώ να μας δώσετε όλες τις δυνατές ενισχύσεις και βοήθειες που είναι διαθέσιμες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι τις χρειαζόμαστε. Θα έλεγα τέλος ότι ανέκαθεν ε, στη Γαλλική οι γυναίκες όντως δούλευαν στη θάλασσα, αλλά συμπληρωματικά, ε, ε, ως συμπληρωματικό εισόδημα για να συμπληρώσουν ούτως ώστε το καλάθι της νοικοκυράς ε, να εμπλουτιστεί με περισσότερα προϊόντα, με περισσότερο ψωμί, περισσότερο γάλα για τα παιδιά κτλ. Χάρη όμως στις δικές μας προσπάθειες, επιτέλους και ευτυχώς, αυτή η δουλειά έχει αναγνωριστεί ως επάγγελμα, δεν θεωρείται πλέον επικουρική, επιπρόσθετη έτσι, εργασία, αλλά πλήρης εργασία, πολύ σημαντική δουλειά δουλειά. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί έτσι αποφεύγουμε καταστάσεις κατά τις οποίες κανείς ε, ε, ε, σκύβει το κεφάλι και δεν ζητά και δεν απαιτεί τα δικαιώματά του. Με τη δική μας ένωση, με τη σε υπόλοιπε οργανώσεις αυτό που προσπαθούμε είναι να κάνουμε τον κλάδο πιο ορατό και να φανεί ο επαγγελματισμός του. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Αυτό είναι ε, βέβαιο και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Κάνια παρακαλώ, έχει τον λόγο. Η σενιόρα Κάνια. Εγώ θα ήθελα να ανταποκριθώ στην απάντηση της ερώτησης που διατυπώθηκε από την Ευρωβουλευτήνα προηγούμενα για τη συνεισφορά μας, τις παρεμβάσεις μας για την κοινή πολιτική αλληλείας. Θα ξεκινούσα λέγοντας ότι υπήρξε πραγματικά μια εμπλοκή και συμμετοχή των ενώσεων και συλλόγων και σε αυτή την περίπτωση των οργανώσεων γυναικών στην Αλία για να ανταποκριθούν στη συζήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το πράσινο βιβλίο για την κοινή πολιτική αλίας Θεωρώ ότι συνέβη αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιθανώς και σε κάποιες άλλες χώρες με ε, άλλο τρόπο. Η Ακτέα θυμάμαι ότι είναι η πρώτη ένωση, η οργάνωση που έθεσε ένα τέτοιο ζήτημα θεμελιώδους σημασίας, μια έλλειψη, μια, ε, ένα κενό στο πράσινο βιβλίο. Εμείς στη δική μας περίπτωση για τις Αζόρες και για την Πορτογαλία συνολικά είχαμε μια παρέμβαση ήταν η κυρία Πατράων Νέβες Ευρωβουλευτής που είχε αναλάβει μια τέτοια παρέμβαση και οι οργανώσεις είχαν ένα ενεργό ρόλο παράλληλα με τη δική της παρέμβαση στη συζήτηση. Αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ακριβώς αυτό λοιπόν. Στο πράσινο βιβλίο, στην κοινή πολιτική αλίας, υπήρχε εδώ θέμα απουσίας ε, κονδυλίων για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ε, αλία που δεν προβλεπόταν, δεν είχε ληφθεί υπόψη. Και τώρα για τα σχόλιά μου, εξού και τα σχόλιά μου και η ανησυχία μου ελήφθη υπόψη αυτό σε σχέση με την πράσινη βίβλο, τότε περνάμε σε μια νέα φάση έχοντας αυτό ληφθεί υπόψη. Πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο της προσοχής το τι θα γίνει σε πραγματικούς όρους στο μέλλον για αυτό το θέμα. Και αυτό συσχετίζεται, πιστεύω, με τις βαθιές ανισότητες όσον αφορά τις γυναίκες. Σε κάποιες από αυτές τις πτυχές αναφερθήκαμε προηγούμενα. Οι γυναίκες, η δουλειά των γυναικών, στο, στον οικοκυριό λέει επικεντρώνεται και στην ε, αλληλεία είναι απλά βοηθητική και η δουλειά στον οικοκυριό πάλι και αυτή δεν αναβαθμίζεται και δεν ε, αναγνωρίζεται, δεν ε, έχει την αναγκαία αναγνώριση. Όλα αυτά λοιπόν που αφορούν τη δουλειά των γυναικών με, αυτές, με αυτές τις αποχρώσεις εξακολουθούν είναι υποτιμημένα. Πρέπει να αναβαθμιστεί αυτή η δουλειά. Η δουλειά είναι αυτή που κάνουν οι ενώσεις των γυναικών για να αναβαθμιστεί η δουλειά των γυναικών στην αλία και να περάσουμε σε ένα μεγαλύτερο, ε, ε, υψηλότερο επίπεδο. Θέλω να τονίσω εδώ ότι σε σχέση με το μέλλον, πέρα από όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν προηγούμενα, από διάφορες παρεμβάσεις ε, και διαφορετικά θεσμικά όργανα εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να είμαστε σε εγρήγορση τι θα γίνει στον τομέα της αλίας. Και για παράλληλα με αυτό και για άλλα θέματα που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη της πολιτικής αλλίας. Το θέμα της ισότητας όμως ανδρών και γυναικών είναι πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Η αξιολόγηση της δουλειάς των γυναικών, η, αναβάθμιση της δουλειάς τους πρέπει να ε, μπορέσει να ε, επιτευχθεί για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα στον τομέα της αλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κάνια. Να θα ήθελα να δώσω το λόγο σε αυτό το σημείο στον κύριο Περέιρα υψηλό αξιωματούχο της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι μπορεί να επεκταθεί επίσης στο θέμα της νέας οδηγίας του 2010 και μπορεί βεβαίως και να απαντήσει στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να παρουσιάσω σύντομα την οδηγία 1041 που υιοθετήθηκε κυρίως χάρη στην υποστήριξη το, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Γυναικών, του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην υιοθέτηση αυτής της οδηγίας. Έγινε πολλής λόγος στις παρεμβάσεις για την έλλειψη αναγνωρισιμότητας και ορατότητας της εργασίας των γυναικών στον τομέα της αλίας αυτό είναι και κάτι που υπάρχει και σε άλλους τομείς. Δεν υπάρχει αποκλειστικά στον τομέα της αλίας. Έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια συζήτηση για την γεωργία και για άλλους τομείς. Και ήταν από τους στόχους αυτής της οδηγίας. Η οδηγία αυτή ε, καταργούσε μια οδηγία του 86. Από το 86 λοιπόν τα κράτη-μέλη ε, είχαν ε, το, την ισότητα μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα ανεξάρτητα επαγγέλματα στις νομοθεσίες τους και την αναγνώριση των, ε, της εργασίας των συζύγων που βοηθούν ή που συνεργάζονται, συνεργάτες όπως λένε στην Γαλλία. Η οδηγία του 86 δεν επέβελε καμία υποχρέωση νομική στα κράτη-μέλη, έκανε μάλλον συστάσεις και δεν επέβαλε υποχρεώσεις δεν έδινε δικαιώματα. Είναι μια οδηγία που δεν μεταφέρθηκε στην νομοθεσία των κρατών μελών και είχε πολύ λίγες πρακτικές επιπτώσεις. Ελπίζουμε και εγώ το ελπίζω και είμαι και πεπισμένος ότι αυτή η οδηγία που υιοθετήσαμε τώρα το 2010 θα αλλάξει την κατάσταση. Πώς αυτό, διότι πρώτα απ' όλα τώρα με αυτήν την οδηγία τα κράτη-μέλη θα έχουν πραγματικές νομικές υποχρεώσεις και όσον αφορά στους συζύγους που βοηθούν, διότι αυτό φορά περισσότερο τα άτομα που είναι εδώ παρόντα, υπάρχει πραγματική υποχρέωση στα κρατημέλη να δώσουν την δυνατότητα στους συζύγους, στις συζύγους που βοηθούν σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην Αλία, να έχουν κοινωνική προστασία όταν υπάρχει κοινωνική προστασία στα κράτη-μέλη για τον ανεξάρτητο, τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι όταν η οδηγία μιλάει για σύζυγο, ε, περιλαμβάνει επίσης ε, και τους συμβίους. Ε, δεν είναι μόνο τα άτομα που έχουν παντρευτεί, είναι κάθε άτομο, κάθε σύντροφος, κάθε συμβίος, συμβία που δεν είναι μισθωτός ε, δεν είναι οικονομικές συνέτερο στην επιχείρηση, εργάζεται τακτικά για την οικογενειακή επιχείρηση. Υπάρχει λοιπόν υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν ούτως ώστε όλα τα άτομα να μπορούν να επωφεληθούν από μια κοινωνική προστασία. Δεν υπάρχει όμως υποχρέωση να καταστεί αυτό υποχρεωτικό. Η οδηγία προβλέπει ότι αυτή η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη μπορεί να γίνει είτε με τρόπο εκούσιο εθελοντικό είτε με τρόπο υποχρεωτικό. Αυτή ήταν, αυτός ήταν ο συμβιβασμός που πετύχαμε στο επίπεδο του Συμβουλίου και αυτό θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη όπου αυτό καθίσταται υποχρεωτικό, όπως είπαμε στην Γαλλία, σε άλλους τομείς και σε άλλες χώρες, να διατηρήσουν την, το καθεστώς, αλλά δεν υπάρχει γενική υποχρέωση για να γίνει αυτό αυτόματα υποχρέωση. Όποιο και αν είναι το σύστημα, ε, το κράτος μέλος ε, έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει αυτήν την ε, δυνατότητα στο νόμο που μεταφέρει την οδηγία και δημιουργώντας αυτήν τη δυνατότητα ρητά στο νόμο θα έχουμε κάτι που δεν είναι μια ρητή υποχρέωση, αλλά που θα είναι έμμεση συνέπεια της οδηγίας. Θα πρέπει να νομοθετήσουμε για το καθεστώς του συμβίου, του συντρόφου που βοηθάει. Διότι έχουμε το άρθρο 5, το άρθρο 7, το άρθρο 8, προσδιορίζοντας τι είναι ο συμβίος, η συμβία που βοηθάει. Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόσωπο που λείπει σε πολλά κράτη-μέλη, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες της οδηγίας, Νομίζω ότι δεν είναι εδώ ε, η κατάλληλη στιγμή. Θα μείνω μέχρι το τέλος και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις, ακόμα και διμερώς αν υπάρχουν ή αν θέλετε ε, να διευκρινίσω. Είμαι στη διάθεσή σας, δεν ξέρω ποιοι είναι οι χρονικοί περιορισμοί. Ευχαριστώ. Ναι, έχουμε καθυστερήσει, λέει η Πρόεδρος. Δεν θέλω όμως ε, να σας στερίζω το δικαίωμα να θέσετε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Σελεστίνη, αναφορικά με την τελευταία παρέμβαση, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι όντως έχει σημασία να αναγνωρίσουμε το καθεστώς του συντρόφου ή του συμβίου. όμως θα πρέπει να υπάρχει ισοτιμία με τους αυτοαπασχολούμενους. Εάν όμως γίνει κάτι τέτοιο, ίσως δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί ε, συχνά είναι ε, πολύ επαχθείς οι κοινωνικές συνεισφορές. Ίσως δεν είναι το κατάλληλο μοντέλο αυτό ε, για την ε, αλληλευτική δραστηριότητα μικρής κλίμακας. Ίσως είναι εξαιρετικά επαχθές κάτι τέτοιο και δίσκαμπτο. Στην Ιταλία καλό θα ήταν να ακολουθήσουμε ένα ειδικό καθεστώς. Ε, συνεισφορές οικογενειακών επιχειρήσεων που να ε, μπορούν να αναλυφθούν πράγματι, δηλαδή να υπάρχει σωστή ε, κοινωνική ασφάλιση, ε, επιδόματα στις γυναίκες και στην οικογένεια. Όμως ε, υπάρχει διαφορετική μεταχείριση συγκριτικά με τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην γεωργία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη της και να εξετάσει πώς θα βελτιώσει την κατάσταση. Οι αλλιευτικές εκμεταλλεύσεις, οι επιχειρήσεις αυτές ίσως δεν είναι τόσο μεγάλες, μεγάλες και δεν μπορούν να καλύψουν, να, ε, ε, να πληρώσουν τις εισφορές που μπορούν να πληρώσουν οι άλλοι. Είναι σαφές, λέει η Πρόεδρος. Θέλει ο κύριος Περέιρα να απαντήσει. Αυτό είναι αρμοδιότητα κράτους μέλους, φαντάζομαι. Αλλά αν θέλετε κάτι να προσθέσετε ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλύτερα να το πείτε εσείς παρά εγώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω τα όσα είπατε. Η Επιτροπή ε, δεν έχει πραγματικά νομική υπόσταση ε, σύμφωνα με τη συνθήκη για να αποφασίσει αυτό που λέτε, δηλαδή ένα ειδικό καθεστώς. Είναι μια αρμοδιότητα που είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό που κάναμε αυτή την οδηγία είναι να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι ελάχιστες συνθήκες που πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη ε, για να υλοποιήσουν την αρχή της ισότητας ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι μια πραγματική αρμοδιότητα κοινοτική. Ως προς την κοινωνική προστασία κάναμε το απαραίτητο για την υλοποίηση της ισότητας μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε λεπτομερώς τα καθεστώτα, τα συστήματα, ε, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση δεν έχουμε καμία νομική αρμοδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, λέει η Πρόεδρο, σημειώνουμε τις, ε, τους προβληματισμούς της κυρίας ε, Σελεστίνη και θα δούμε ποια συνέχεια θα δώσουμε σε αυτό το θέμα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν το πρώτο μέρος της ακρόασης αυτής. Ε, έχουμε κάπως καθυστερήσει, ωστόσο πιστεύω ότι άξιζε το κόπο να ακούσουμε την άποψη όλων. Το δεύτερο μέρος της ακρόασης έχει να κάνει με την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΦΕΠ και τον ρόλο των διαχειριστικών αρχών ή των διαμεσολαβητών και των τοπικών ομάδων δράσης. Να δώσω το λόγο καταρχάς στην κυρία Μόνικα Μπούρχ του της μονάδας στήριξης FARNET που είναι το δίκτυο ε, ζωνών αλλία στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας ε, να πάρω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής σας. Με λένε Μόνικα Μπέρτς από την Μονάδα Στήριξης του Φάρνετ. Εμείς προσφέρουμε συμβουλευτική στήριξη στη Γενική Διεύθυνση για τις Αλληλευτικές Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στηρίζουμε επίσης τις διαχειριστικές αρχές και τα τοπικά, τις τοπικές ομάδες δράσης για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Ελπίζω με την παρουσίασή μου σήμερα να σας ενθαρρύνω να αξιοποιήσετε όλες αυτές τις ευκαιρίες, να έχετε πρόσβαση σε κονδύλια για να καλύψετε πολλές από τις ανάγκες που έχετε ε, επισημάνει. Να σας εξηγήσω τι είναι ο άξονας 4. Ε, ποιες είναι οι τοπικές ομάδες δράσης για την αλληλεία, τις οποίες ονομάζουμε FLAG. Στη συνέχεια θα μιλήσω για το δυναμικό που κρύβεται πίσω από αυτά τα εργαλεία και πίσω από αυτές τις δυνατότητες, ε, κάτι που μπορούν να αξιοποιήσουν οι γυναίκες. Και στο τέλος θα παρουσιάσω κάποιες από τις ιδέες που έχουν ήδη προκύψει, κάποια από τα πορίσματα από τη δουλειά των τοπικών ομάδων δράσης για την αλία. Και θα παρουσιάσω και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ε, για το οποίο θα μπω σε λεπτομέρειες. Ποιος είναι ο άξονας 4 λοιπόν. Είναι ένας άξονας προτεραιότητας ε, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας. Είναι ένας καινούριος άξονας για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Για πρώτη φορά λοιπόν γίνεται προσπάθεια να ε, λυθούν κάποια από τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, δηλαδή διατήρηση αποθεμάτων, μείωση, ε, επίλυση του θέματος της μείωσης της κερδοφορίας μεταξύ άλλων. Έχουμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κάθε κλάδος εξετάζονται στο πλαίσιο της περιοχής όπου σημειώνονται. Ε, εάν πρόκειται για μια εξόχως απόκεντρη περιοχή ή μια αλλιευτική περιοχή στη Μεσόγειο, όπου δυσκολεύεται ο αλλιευτικός κλάδος να ανταγωνιστεί τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισμός ή η υπερβολική αστικοποίηση της παράκτειας περιοχής και ούτω καθεξής. Επομένως, με τον άξονα 4 έχει αλλάξει πλέον, έχει σημειωθεί μια μεταστροφή του παραδείγματος στην ευρωπαϊκή πολιτική για την αλία, γιατί στόχος πλέον είναι συγκεκριμένες προτεραιότητες. Έχουν εντοπιστεί τομείς που χρειάζονται περιοτεραιότητα. Είτε πρόκειται για αλλιευτικές κοινότητες, είτε πρόκειται για κάτι άλλο. Τα κονδύλια λοιπόν ε, τα αξιοποιούν οι τοπικές ομάδες δράσης με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε περιοχής. Ε, υπάρχει στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και γι' αυτό η προσέγγιση είναι πάντοτε από κάτω προς τα πάνω. Στόχος μας είναι ε, να αποφύγουμε αυτή τη θηρίδα της επικράτειας, της εκάστοτε, αυτό το οποίο στα γαλλικά λέγεται territoire guichet, και να πάμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε territoire projet και όχι γκισέ. Να ε, μην είναι μια θηρίδα, δηλαδή ένα γκισέ που κατανέμει τα κονδύλια, αλλά να έχουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο για το μέλλον. Ε, τι θέλουμε να πετύχουμε, ποιο είναι ο καλύτερο τομέα για να δράσουμε, πώ θα τα καταφέρουμε όλα αυτά. Να υπάρχει ένα σχέδιο δηλαδή. Υπ' αυτή την έννοια ε, τα κονδύλια του άξονα 4 βεβαίως και στοχεύουν στις γυναίκες. Είναι ευκαιρία για τις γυναίκες να συμμετάσχουν στις ε, τοπικές ομάδες δράσης για την αλία. Μπορούν έτσι να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση και χάραξη της στρατηγικής και να κινήσουν τα πράγματα προς την κατεύθυνση που επιθυμούν προκειμένου να βελτιώσουν και τη δική τους προσωπική κατάσταση. Πέρα από όλα αυτά, οι γυναίκες ούτως ή άλλως είναι το 50% του πληθυσμού στον οποίο στοχεύουμε και χαρακτηρίζονται από δυναμικότητα πάρα πολύ συχνά. Είναι ένα πολύ καινούριο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον άξονα υπαριθμών 4. Ε, χρειάζεται δουλειά, γιατί όποιος υποβάλλει πρόταση θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη ε, στρατηγική ανάπτυξη. Είναι δύσκολο να αλλάξει η νοοτροπία και ξέρουμε ότι οι γυναίκες είναι εξαιρετικά ανοιχτές, έχουν ένα ανοιχτό πνεύμα. Ίσως επειδή ε, το τρέχον σύστημα της κρατά αρκετά στο περιθώριο, ε, ψάχνουν την παραμικρή ευκαιρία για να βελτιώσουν τη θέση τους και αυτό είναι πολύ θετικό. Ε, και ίσως επειδή το σύστημα της κρατά στο περιθώριο έχουν αυτή τη στιγμή λιγότερα συμφέροντα και λιγότερα πράγματα να χάσουν με τις αλλαγές. Βλέπετε τον κατάλογο των μελών. Έχουμε διαφοροποίηση πολύ ισχυρή και οι γυναίκες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτό. Και έχουμε και τις συνδέσεις στον ίδιο τομέα, από την παραγωγή μέχρι τις πωλήσει και την διανομή, αλλά και τις συνδέσεις με άλλους τομείς, συνδέσεις με το τουρισμό για παράδειγμα. όπου και εκεί ε, οι γυναίκες δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Να πάρουμε τώρα μια γεύση για, το, για τα ποσά για τα οποία μιλάμε. 21 χώρες ε, εφήρμοσαν και ε, τον άξονα υπαριθμών 4. 13% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας. Διαφορετικός προϋπολογισμός, τελείως διαφορετικά νούμερα από τη μία χώρα στην άλλη, όπως βλέπετε στη διαφάνεια και έχουμε προϋπολογισμό από 1 εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο της προγραμματικής περίοδου στην Κύπρο μέχρι και 234 εκατομμύρια ευρώ στην Πολωνία. 234 φορές περισσότερο. Και με την Εθνική συγχρηματοδότηση συνολικά ε, φτάνουμε στα 826 εκατομμύρια ευρώ δημοσίων επενδύσεων, επενδύσεων από δημόσιους φορείς, είτε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τις κρατικές αρχές. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από ό,τι είχαμε φανταστεί, γιατί είναι ένα καινούριο πρόγραμμα και ε, θα έπρεπε πρώτα να καταρτιστούν οι ενδιαφερόμενοι και να αποκτήσουν τις κατάλληλες ε, δεξιότητες και δυνατότητες. 169 τοπικές ομάδες δράσης για την αλία έχουν ήδη δημιουργηθεί και ελπίζουμε το νούμερο αυτό να φτάσει στις 250 μέχρι την επόμενη χρονιά. 3 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός πάνω κάτω ανατοπική ομάδα δράσης για την αλία. Βεβαίω ε, τα επίπεδα προϋπολογισμού διαφέρουν τα ομάλα από τη μία τοπική ομάδα δράση στην άλλη. Αυτό το αριθμιστικό στοιχείο αποτελεί ένα μέσο όρο. Στην Ισπανία βλέπετε ότι είναι 3 ε, εκατομμύρια, αλλά γιατί, γιατί έχουμε από λιγότερο από 1 εκατομμύριο μέχρι και 10 εκατομμύρια στην εσωτερική κατανομή στην χώρα αυτή. Τώρα, τι είδους προγράμματα χρηματοδοτεί ο άξονας υπαριθμών 4. Ε, εξαρτάται αυτό από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από 1 εκατομμύριο μέχρι 60 εκατομμύρια στην Πολωνία. Αναλόγως με τα ισχυρά σημεία, τις αδυναμίες ε, σε κάθε τομέα. Ε, εξαρτάται και από το μέγεθος του αλλιευτικού ε, κλάδου. Πολύ συχνά είμαστε στο 5% ή αλλού στο 15%. Άρα η δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων είναι τεράστια πρόκληση. Εάν κανείς, ας πούμε, μπορεί να αξιοποιήσει 50 εκατομμύρια και η αλληλής είναι μόνο 15, είναι κάπως δύσκολο να αξιοποιήσει το σύνολο των κονδυλίων μικρά πιλωτικά προγράμματα υλοποιούνται και εφαρμόζονται εκεί που ο προπολογισμό δεν είναι υψηλό. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε υψηλό προπολογισμό, θα μπορούσαν να γίνουν μόνο μελέτε ή δραστηριότητε αδελφοποίηση περιοχών, ε, στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προγράμματα ευρείας ε, διαφοροποίησης. Να, να σας δώσω μια γενική ιδέα για τις ιδέες που ε, βρισκόμαστε στην αρχή των προγραμμάτων και των συζητήσεων για να ξεκινήσουν όλα αυτά και ένας κατάλογος των μέτρων για τις δυνατότητες και την πρόσβαση. Μέχρι στιγμής η διαχείριση αυτών των πρωτοβουλειών σε σχέση με την δυνατότητα παροχής στις οργανώσεις γυναικών στον τομέα των, της Αλίας και στην Ανδαλουσία και στις Αστούρης και στην ε, ε, Γαλλικία και βλέποντας υπόψη τα θέματα τα οποία η Νατάλια είχε αναφέρει και για άλλες περιοχές δυνατότητες πρόσβασης σε κονδύλια και υποστήριξη στις δικές τους περιοχές πρόσβαση σε σχέση με την κατάρτιση και υποστήριξη επιμόρφωσης γυναικών. Και τέλος, χρηματοδοτική υποστήριξη για συγκεκριμένα εξειδικευμένα προγράμματα που είναι στα χέρια των γυναικών ή που τα ε, διαχειρίζονται γυναίκες και δουλεύουν και εργάζονται για γυναίκες ε, προωθώντας τις δραστηριότητες των γυναικών στον τομέα της αλληλείας αλλά και των προϊόντων τους ε, ώστε να υπάρξει πρόσθετη αξία που θα απορρέει σε σχέση με αυτά τα προϊόντα. Προγράμματα για τον τουρισμό, βελτίωση των όρων εργασίας επίσης καθώς και η ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών προστασία και περίθαψη για τους ηλικιωμένους ε, που όχι μόνο δημιουργεί θέσεις απασχόλησης αλλά και μέσα από αυτή τη δραστηριότητα δίνει τη, δίνονται δυνατότητες να είναι πιο ευέλικτες οι γυναίκες σε σχέση με την εργασία τους. Τέλος θα ολοκληρώσω με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την Ισπανία που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Είναι οι εξορρυκτικές δραστηριότητες ε, ε, γυναικών και σε αυτό το πρόγραμμα έχει επεκταθεί το πλαίσιο σε διαφορετικές δραστηριότητες που αποτελούν μέρος του συνόλου που ε, αφορούν τα οστρακόθερμα και τη συλλογή τους, διευρύνοντας τις δραστηριότητες από την εξορρυκτική δράση, δραστηριότητα στην μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων αυτών κάποιος αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα προηγούμενα αυτό, απορρέει από την ε, ε, αγορά ενός ε, μιας συσκευής καθαρισμού ώστε να μπορούν να περνούν τα προϊόντα τους στην αγορά με την αγορά ακριβώς ενός τέτοιου εξοπλισμού μπορούν οι γυναίκες τώρα να πωλήσουν τα προϊόντα τους και έχουν υποστηριχθεί στην ανάπτυξη επαφών με αγοραστές και ε, συνειδητοποιώντας ε, οι αγοραστές ε, την ποιότητα των προϊόντων τους να μπορέσουν να βρουν δυνατότητες σε τοπικά ξενοδοχεία και εστιατόρια που δίνουν παραγγελίες και έτσι βλέπουμε ότι αυτό συμπληρώνεται και με ξεναγήσεις, ξεναγήσεις για τουρίστες ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν αυτές τις δραστηριότητες ε, επισκεπτόμενοι τις περιοχές αυτές, ε, τουρίστες και να γνωρίσουν και τα προϊόντα. Βλέπουμε και τη δυνατότητα γεύση γνωστικών ε, τέτοιων εμπειριών, καθώς επίσης και δυνατότητες για να αποκτήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό, συνταγές για την να μπορούν να μαγειρεύουν αυτά τα προϊόντα, ε, τη δυνατότητα να ε, δημιουργούν ε, και καλάθια. Όλα αυτά δίνουν μια ευρεία εικόνα. Είναι ένα παράδειγμα βέβαια αυτό ενός συγκεκριμένου προγράμματος όπου άνδρας, άνδρες ή γυναίκες έχουν αναλάβει δραστήριο ρόλο για να βελτιώσουν τη ζωή τους ε, εμπλεκόμενοι περισσότερο σε σχέση με το κοινωνικό έργο και τις κοινωνικές σχέσεις προσθέτοντας ε, ε, πρόσθετη αξία ή αναβαθμίζοντας την εργασία τους σε σχέση με τις δραστηριότητε τους και την, τις σχέσεις με την τοπική τους κοινωνία. Αυτά είναι και στα θέματα γευσηγνωσίας, δημιουργίας καλαθιών που πλέκουν με την δυνατότητα ε, να έχουν την ε, διάθεση των προϊόντων τους. Δράτω με τις ε, για να αναφέρω ακόμα και το link για την ομάδα εργασίας και συζητήσεων που έχουμε. Στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Προσβλέπουμε στο να υποβληθούν ιδέες, προτάσεις, πληροφορίες από εσά μεταξύ ημών και ατόμων που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα ε, γυναικών προτείνοντας ε, σχέδια ε, για διαδικτύωση και συνεργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μόνικα Μπρόκη για αυτές τις πληροφορίες και για να μπορέσουν αυτά να ληφθούν υπόψη και περνάμε στον τελευταίο που θα παρέμβει που είναι ο κύριος Χωσέ Λουίς Γκονθάλες Σεράνο που θα μας παρουσιάσει ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε πρόσφατα και που έχει τον τίτλο Ισπανικό Δίκτυο Γυναικών στον τομέα Λίας. Είναι ο Γενικός ε, Διευθυντής ε, από πλευρά της Γενικής ε, Γραμματείας για τα θαλάσσια θέματα όσον αφορά την υπηρεσία στο Υπουργείο του και ο κύριος Γκονθάρες Θεράνο έχει τον λόγο. Παρακαλώ σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ φυσικά για την ευκαιρία που μας δίνεται από την Επιτροπή να παρουσιάσουμε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή. Θα σας μιλήσω αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία ενός δικτύου γυναικών στον αλλιευτικό τομέα που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Ο Ισπανικός τομέας της Αλίας, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένας τομέας πραγματικά ευρύτατος φαίνεται σε σχέση με τις διαφάνειες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας ε, τώρα εδώ μπροστά μας. Έλεγα ότι ο Ισπανικός ε, τομέας αλληλείας είναι ευρύτατος. Οι γυναίκες εκπροσωπούνται σε κάθε ένα από τους υποτομείς. Η σημασία που έχουν ε, συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της κάθε δραστηριότητας. Δεν είναι τα ίδια τα, στον εξορρυκτικό ε, τομέα των οστρακοδέρμων, όπου οι γυναίκες έχουν ε, ένα ποσοστό 17% με άλλους τομείς που παραδοσιακά είναι παραδοσιακά γυναικοί τομείς όπως σε σχέση με τον, την ε, επισκευή δικτύων, τη συσκευασία ή την ε, εξορρυκτική δραστηριότητα των που αφορούν την τοποθέτηση των αλλιευμάτων μέχρι το μαγαζί που ε, θα απολυθούν, όπου η παρουσία και συμμετοχή της ε, γυναίκας είναι πλειοψηφική, όπως και στην μεταποίηση με ένα 75% της συμμετοχής γυναικών, όπως επίσης και στην υδατοκαλλιέργεια με 45% και αντίστοιχα ποσοστά. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ταυτοποιούν και δίνουν την εικόνα της γυναίκας στον αλληλευτικό τομέα στην Ισπανία. Ποια προβλήματα μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ως κυριότερα προβλήματα. Έχουμε κάποια κοινά σημεία σε σχέση με τον ανδρικό τομέα, όπως για παράδειγμα η απουσία ε, κατάρτισης, ε, επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είναι η, εργασ... η εργασίας ε, ή όπως είναι τα ε, προβλήματα της ε, αλλαγής των γενεών αλλά και πιο χαρακτηριστικά και εξειδικευμένα προβλήματα σε σχέση με την απασχόληση των γυναικών από την άλλη πλευρά, όπως είναι η αναγνώριση του επαγγελματός τους ε, που συνδέεται άμεσα με την δυνατότητα να μπορέσουν να αναβαθμιστούν οι δραστηριότητές τους, αλλά επίσης ε, και τον ευάλωτο χαρακτήρα της εργασίας τους. Ε, έχουμε κάποια στοιχεία που τεκμηριώνουν όλα αυτά. Έχουμε κάποια λίγα στοιχεία. Είναι αναγκαίο λοιπόν να συλλέξουμε και να έχουμε μια τράπεζα δεδομένων για αυτά τα στοιχεία. Όσον αφορά την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των ε, γυναικών, των δραστηριοτήτων των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Ταμείο των, για την Αλία δεν αναγνωρίζει τη δραστηριότητα των, της εξορρυκτικής ε, ε, δραστηριότητας για τα οστρακόδερμα δεν αποτελούν ένα εξειδικευμένο επάγγελμα, δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό τμήμα. Επιθυμούμε όλοι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο να αναγνωριστούν ε, οι εξορρυκτικές αυτές δραστηριότητες, η συσκευασία, επίσης η δραστηριότητα συσκευασίας των προϊόντων ως ξεχωριστό επάγγελμα. Όσον αφορά τώρα την ε, επαγγελματική, ε, ας το πω έτσι, σταθερότητα, αντιμετώπιση του ευάλωτου χαρακτήρα θα πρέπει να δούμε ποιες ήταν οι επιπτώσεις όλων των ενισχύσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέχρι σήμερα στα διαφορετικά λιμάνια της Ισπανίας. Όπως ε, για παράδειγμα στο Βίγο, όπου τα τελευταία δέκα χρόνια είδαμε πώς μειώθηκε η απασχόληση σχετικά. Για την μείωση αυτή της απασχόλησης οι πρώτοι που πλήττονται είναι οι γυναίκες βέβαια το 2000 η απασχόληση των γυναικών ήταν 9%. Από το 2009 μόνο 6,6%. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μειώθηκε κατά 44% η απασχόληση στο λιμάνι του Βίγο ένα 59% κατά μέσο όρο κατά μέσο όρο μειώθηκε για τις γυναίκες όμως. Βρισκόμαστε εν ώψη μιας ε, κοινωνικής ιδιομορφίας αυτής της δουλειάς ε, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτου του χαρακτήρα και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο με προτεραιότητα της κοινωνικής πολιτικής. Όχι τη μόνη προτεραιότητα, φυσικά έχουμε και άλλες προτεραιότητες στην ε, κοινωνική πολιτική. Τα θέματα των ζωνών που εξαρτώνται από την αλληλεία, παράκτιων ζωνών, των ε, διαφόρων ε, ε, εργαζομένων στα σκάφη καθώς επίσης και των μεταναστών και προερχόμενων από τρίτες χώρες που εργάζονται στα σκάφη που ψαρεύουν στην ανοιχτή θάλασσα και να υπάρξουν όλα τα στοιχεία σχετικά και άλλα θέματα για την κοινωνική πολιτική. Αλλά η πολιτική για την ισότητα των γυναικών πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητές μας και σε αυτό ακριβώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να εργαστούμε. Πώς να αντιμετωπιστούν τώρα όλα αυτά τα προβλήματα. Η εργασία των γυναικών και επανειλημμένα το είπαμε αυτό σήμερα το απόγευμα είναι μια αόρατη θα έλεγα εντό εισαγωγικών εργασία για μια ολόκληρη ε, σειρά λόγων που ε, η ίδια η παράδοση κάνει τις γυναίκες να μην έχουν διάκριτο χαρακτήρα και για να μπορέσουμε να διαρρήξουμε αυτό το φαύλο κύκλο των παραδοσιακών αξιών και της παράδοσης πρέπει να ε, μπορέσει να ενεργοποιηθεί η γυναίκα και να ε, μπορέσει να δραστηριοποιηθεί σε ενώσεις συλλόγους τότε αποκτά δύναμη τότε μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στη ζωή της. Και αυτή είναι ακριβώς η στιγμή τώρα όπου η διαδικτύωση αρχίζει να δικαιολογείται και αρχίζει να είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη. Στην Ισπανία έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν είναι ίδιες οι προϋποθέσεις και οι όροι ε, παντού στην Ισπανία, αλλά έχουμε σε κάποιες περιοχές αυτές τις δυνατότητες, όρους και προϋποθέσεις να ενεργοποιηθούν οι γυναίκες και να ενταχθούν σε δίκτυα ενώσεις συλλόγου. Είναι καλή λοιπόν ιδέα να δραχθεί κανείς ε, του άξονα αυτού της ε, δυνατότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας ε, για να δραστηριοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο. Αυτή η δυνατότητα θα ήταν να ενταχθεί ακριβώς στον κανονισμό για την αλληλεία αυτό και να προβλέπεται ώστε να καλύπτεται αυτή η ανάγκη Μα έδωσε τη δυνατότητα να αναλάβουμε πρωτοβουλία, εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο. Ένα δίκτυο το οποίο στήχησε, κόστισε πολλές προσπάθειες, έγινε όμως πραγματικότητα στην, κατά την έναρξη του 2010. Πρέπει όμως ε, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα ακόμα και πρέπει να πείσουμε ότι το να συνεχίσουμε προάγοντας τους στόχους της ισότητας όχι μόνο θα πρέπει να είναι δεκάρικοι λόγοι που θα ακούγονται αλλά πρέπει να αποκτήσουν όλα αυτά σάρκα και οστά. Και αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε από τη Γενική Διεύθυνση για τις θαλάσσιες υποθέσεις ε, να προαγάγουμε αυτά τα θέματα δημιουργία ενός δικτύου ακριβώς ε, για την αλληλεία για τις γυναίκες. Το πιο σημαντικό εφέτος τι ήταν. Ήταν ακριβώς ε, η διάχυση των στοιχείων αυτών στο, αυτού του δικτύου, ο ευδιάκριτος χαρακτήρας που θα αποκτούσαν αυτές οι δραστηριότητες. Καταφέραμε μέσα σε ένα χρόνο να έχουμε μία σελίδα στο ε, διαδίκτυο για τις ε, δράσεις αυτές που στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλλιές μια ολόκληρη σειρά εγχειριδίων και μαθημάτων, αγγλικά, πληροφορική, επιπλέον μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή εμπειριών και την ε, ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο. Πέρα από αυτά το πιο σημαντικό όμως είναι για αυτή την περίοδο στην οποία αναφέρομαι η προσπάθεια που έγινε να πάμε εκτός Μαδρίτης ε, και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο για να καταφέρουμε να ε, συλλέξουμε, να προσελκύσουμε κόσμο σε σχέση με αυτή τη διαδικτυακή ε, δραστηριότητα. Με μια ολόκληρη σειρά σεμιναρίων, εκδηλώσεων, με τη διεξαγωγή του πρώτου συνεδρίου, του πρώτου κογκρέσου που μας έδωσε την ευκαιρία εφέτος ε, να παγιώσουμε τη θέση μας ως δίκτυο. Και σε σχέση και με την κυβέρνηση της χώρας των Βάσκων στο Σαν Σεμπαστιάν, καταφέραμε να προσέθουν σε αυτό το συνέδριο πάνω από 350 συμμετέχοντες. Συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το δίκτυο ΑΚΤΕΑ, από την Λατινική Αμερική, καθώς επίσης και από πολλές ενώσεις και συλλόγους ε, από την Ισπανία. Τι, θέλουμε να κάνουμε, τι θέλαμε να κάνουμε με αυτό το συνέδριο. Να δώσουμε ευδιάκριτο, ορατό χαρακτήρα και ρόλο στις δραστηριότητες αυτές των γυναικών. Να εμβαθύνουμε στην ε, δραστηριότητα στις ενώσεις αυτές ε, των γυναικών, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει παραπέρα το κίνημα διεκδικήσεων τους. Ε, γιατί αν παραμέναμε ε, στάσιμοι δεν θα μπορούσαμε να πάμε πιο πέρα και να πετύχουμε κάτι παραπάνω. Για να ολοκληρώσω δύο λόγια μόνο για το μέλλον αυτού του δικτύου δεν θα μακρηγορήσω. Αν θέλετε να διατυπώσετε μια ερώτηση στη συνέχεια, είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω. Τι θα κάνουμε του χρόνου, 2011, που θα είναι χρόνος κλειδί. Θα δουλέψουμε προφανώς για να προχωρήσει η δουλειά αυτή του δικτύου. Θα πρέπει πολλά να γίνουν, θα πρέπει να καταλήξουμε στο να έχουμε πάνω από χίλια μέλη στο δίκτυο, αλλά θα πρέπει επίσης ε, να συνεχίσουμε τις αποστολές ε, σε διάφορες πόλεις ε, και περιοχές για να γνωστοποιηθεί το έργο μας. Σημαντικό όμω είναι να έχουμε μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Για μένα υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές σε αυτή τη στρατηγική. Η πρώτη αναφέρεται στις διεκδικήσεις των γυναικών σε αυτή την περίοδο. Σήμερα ήδη διάφορες τέτοιες διεκδικήσεις σε τίματα αναφέρθηκαν για την, τα κοινωνικά ζητήματα, για τον ευδιάκριτο χαρακτήρα των, της εργασίας τους. Αυτές όμως οι διεκδικήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο αν υπάρχει και η συνιστόσα αυτή για την ισότητα των γυναικών. Καμία από τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα αυτά δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις ε, που διαφοροποιούν τα πράγματα. Θα πρέπει έτσι λοιπόν οι γυναίκες να καταβάλουν προσπάθειες αν θέλουν αυτά τα αιτήματά τους και οι διεκδικήσεις τους να ευδοκιμήσουν. Θα πρέπει σε πραγματικό χρόνο να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αυτά. Ένα μέρος της εργασίας ε, εφ' θα αφιερωθεί να γίνει μια μελέτη, όχι μια θεωρητική μελέτη, αλλά μια πρακτική εξειδικευμένη μελέτη εντοπισμού των προβλημάτων ταυτοποίησης ε, και ε, ιεράρχησης των προβλημάτων. Και για μένα θεμελιώδες θέμα ε, είναι το πιο σημαντικό μέρος της εργασίας μας είναι εκείνο που θα δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε ένα θετικό περίγυρο, καλό κλίμα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τα προγράμματα αυτά για την επιχειρηματικότητα των γυναικών. Σήμερα υπάρχουν κονδύλια ε, για να γίνει κάτι αλλά αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι τα καλά προγράμματα και σχέδια. Αν δημιουργήσουμε όμως ένα θετικό περίγυρο, ένα θετικό κλίμα, όπου αυτές οι ιδέες θα μπορέσουν να ευδοκιμήσουν εκείνα τα άτομα όταν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κάποια ιδέα που μπορεί να μεταφραστεί σε ένα πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να προαχθεί, ε, τότε θα έχουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, θα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού που θα είναι θετικά στοιχεία για να προαχθούν όλα αυτά και να μπορέσει να ευδοκιμήσει, να αναβαθμιστεί η δουλειά των γυναικών. Αυτά είναι όλα όσα ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μην σας κούρασα μετά όσα είπα. No, creo que ha sido muy interesante. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση πιστεύω. Και έτσι ολοκληρώσαμε με τις παρεμβάσεις ε, και μπορούμε αν επιθυμείτε να έχουμε τις ερωτήσεις ή τις παρεμβάσεις για να συζητήσουμε κάποια πράγματα που σας ενδιαφέρουν. La señora Celestini ha pedido la palabra. Ehm, chiedo scusa, è tutto molto giusto quello che ha detto il Όλα αυτά πολύ σωστά τα οποία μας αναφέρατε αυτά τα οποία ο εκπρόσωπος του Ισπανικού Δικτύου ανέφερε. Έχω όμως μια ερώτηση. Γιατί πρέπει εδώ ένας άντρα να μας εκθέσει για τα προβλήματα των γυναικών και την κατάσταση των γυναικών στην Ισπανία. Γιατί ένας άντρα και όχι μια γυναίκα. Ε, Είναι δική μου έμπνευση σε αυτό το πρόγραμμα, αυτό το εγχείρημα. Δική μου έμπνευση προσωπικά. Εδώ και πέντε χρόνια το συνέλαβα, το προχώρησα και όταν θα έχει ολοκληρωθεί θα δώσω τη θέση μου σε άλλο άτομο που θα είναι μια γυναίκα για να δώσει συνέχεια. Ε, Και οι άντρες συνεργαζόμενοι με τις γυναίκες ε, βλέπουμε ότι επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα. υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον και εργάστηκε με, μεγάλο, με μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για να ευδοκιμήσει αυτό το θέμα και το αναγνωρίζουμε αυτό. Κάποια άλλη παρέμβαση υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση θα δώσω τον λόγο στην κυρία Άντρες Μπαρέα που όπως είπαμε είναι μέλος της ε, ε, δικής μας επιτροπής που έχει υπομειστεί. Τι συμβαίνει, λέει η Πρόεδρος, διακόπτη, χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση, δεν ακούγεται. Στην κυρία Άντρες Μπαρέα θα δώσουμε τον λόγο, που έχει αναλάβει την πτυχή της ισότητας ε, για τις γυναίκες. Θα της δώσω τον λόγο για να ολοκληρώσει πρωτού ε, ολοκληρώσουμε εμείς τις εργασίες μας. Πολύ καλά σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους. Η αλήθεια είναι ότι για τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτό το κοινοβούλιο να καταλήξουμε να έχουμε μία ε, ακρόαση ε, υπό ε, όρους και προϋποθέσεις και με μια αίθουσα επαρκώς πλήρη είναι ενδιαφέρον το εγχείρημα και τώρα θα ήθελα να πω ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία σημείωσα και ε, ε, ε, είδα. Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να μου αναφέρετε ως έλλειψη σε σχέση με την παρέμβασή μου να μου το επισημάνετε. Θα ήθελα επίσης η γραμματεία να σημειώσει σε σχέση με τα συμπεράσματα τα οποία θα διανεμηθούν υστερότερα σε μία εβδομάδα σε όσους ενδιαφέρονται. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ταυτοποιήσω κάποια συμπεράσματα. Απόλυτη ανάγκη που υπάρχει να έχουμε στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα που θα μας δίνουν μια πραγματική εικόνα για τον αριθμό των γυναικών, για τους τομείς ανατομέα και για την ποιότητα αυτών των στοιχείων ανατομέα. Είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη των στοιχείων για την ποιότητα. Δεύτερο, το, δεύτερο θέμα, η προσπελασιμότητα στην κατάρτιση, εκπαίδευση τοπικά και εθνικά και περιφερειακά και ευρωπαϊκά, τονίζοντας αυτή την πτυχή και τα εναλλακτικά προγράμματα όσον αφορά την κατάτηση και εκπαίδευση, όπως είναι η δημιουργία μαθημάτων, courses που θα δημιουργούν διάφορες ε, δυνατότητες γευσηγνωσίας, ε, τουρισμού, ξεναγήσεων κτλ. Τρίτη προτεραιότητα, ένταξη της συνιστώσας της παραμέτρου της ισότητας των γυναικών σε όλες τις πολιτικές και προγράμματα. Λόγω της απουσίας των γυναικών και του αόρατου χαρακτήρα των γυναικών της δουλειάς τους. Δύο ή τρεις μόνο εκπρόσωποι βρίσκονται γυναίκες στα ρακ, στα ρακ αυτά και αυτά τα άτομα θα μπορούσαν να μπορέσουν να δράσουν ώστε να υπάρξουν κοινωνικά, κοινωνικά μέτρα αλλά και περιβαλλοντικά μέτρα κοινωνικά το τονίζω σε σχέση με όσους παρενέβησαν, που είναι πολύ σημαντικά, μια και η γυναίκα αποτελεί τμήμα του τομέα της αλληλείας που πολλά αφορούν τα από τα θέματα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Και η οδηγία 86 86-603 με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και τονίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η γυναίκα ως σύζυγος, η γυναίκα ως εταίρος, ως συνεργάτης. Πρέπει να εξειδικευτούν όλα πολύ περισσότερο και σε σχέση και με την κυρία Σελεστίνη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιες χώρες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Να βελτιωθεί η εμπορία, η διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων. Σημαντικό θέμα αυτό το οποίο καθορίζεται ως στοιχείο για να έχουν οι γυναίκες αξιοπρεπή ζωή και αξιοπρεπές εισόδημα, αξιοπρεπή μισθό. Έτσι λοιπόν λοιπόν θα πρέπει και αυτό σημαντικό στοιχείο να αντιμετωπιστεί. Δεν μιλήσαμε πολύ γι' αυτό, αλλά θεωρώ ότι βρίσκεται κάτω και παράλληλα με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και συνοδεύει όλα αυτά η βιοτεχνική αλληλεία στην οποία είναι παρούσα η γυναίκα όπως είπαμε και πιο πριν να μπορεί να έχει πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλληλεία μέσω των flags ή μέσω των αξώνων του, Ταμείου αυτού, γνωρίζοντας τις συγκεκριμένες ανάγκες ε, των γυναικών αυτών. Οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το Ταμείο Αλληλείας και στη μελλοντική μεταρρύθμιση της κοινή πολιτικής Αλληλείας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση, στην ε, βιοτεχνική αλληλεία και στις γυναίκες, στην γυναίκα ως σημαντικό παράγοντα αυτής της παραδοσιακής αλίας. Και ως παράδειγμα αναφέρθηκε αυτό το οποίο ανέφεραν οι παρεμβαίνουσες σήμερα, να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των γυναικών. Και αναφέρθηκε ότι πίσω από κάθε σκάφος, πίσω από κάθε πλοίο υπάρχει και μια γυναίκα και από τα όσα είπε ο κύριος Γκονθάλεθ ότι πρέπει να ξεπεράσουμε συγκεκριμένους φραγμούς και προσκόμματα και εμπόδια. Εμείς είμαστε μέρος του μισού κόσμου, είμαστε ο μισός κόσμος οι γυναίκες ε, της γης και έτσι λοιπόν εμείς οι γυναίκες θα πρέπει σε όλους τους τομείς και στον τομέα τον αλλιευτικό να ληφθούμε υπόψη όπως πρέπει. Η αξία των γυναικών και της δουλειά τους στον τομέα της αλληλείας. Αν κάτι δεν έχω συμπεριλάβει θα ήθελα να μου το αναφέρετε για να ληφθεί υπόψη και η Γραμματεία δεσμεύεται να εκπονήσει ένα κατάλογο των συμπερασμάτων που θα διαβιβαστούν στις εισηγήτριες και στις ενώσεις που δεν παρενέβησαν αλλά είναι εδώ παρόν, παρούσες για να δουν τα αποτελέσματα αυτής της ημερίδας ποια ήταν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εγώ εξ ονόματος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σας ευχαριστώ όλους σας, γυναίκες και άνδρες, για τις παρεμβάσεις σας, για το ότι είσαστε παρούσες σε αυτή την ακρόαση που πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για όλους εμάς που συμμετείχαμε. Η κυρία Άνδρες Μπαρέα, επειδή αναφέρθηκε πιο πριν ότι δεν υπήρχαν επαρκείς βουλευτές για μια τόσο σημαντική ε, ακρόαση σαν αυτή που είχαμε, και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα μέλη της που δεν υπήρχαν επαρκή μέλη να σας ακούσουν και να σας προσέξουν. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από τα συμπεράσματα τα οποία διατύπωσε η εκπρόσωπός μας, να είσαστε βέβαιοι και βέβαιες ότι θα διανεμηθούν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, οι παρεμβάσεις και θα υπάρχουν ε, σε γραπτό κείμενο όλα αυτά διαθέσιμα και εν πάση περιπτώσει θα είναι μια καλή τεκμηρίωση αυτή που θα έχουμε στη διάθεσή μας για το μέλλον και για να συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε τον ρόλο των γυναικών στην αλληλεία. Πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος των γυναικών στην αλληλεία θα πρέπει να μας κάνει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας. Δική μας είναι η μάχη αυτή, ο αγώνας αυτός. Είδαμε πόσο μας δυσκόλεψε τη ζωή, στο παρελθόν μας δυσκόλεψαν τη ζωή κάποια πράγματα. Ο ρόλος <clears throat> θα πρέπει να πούμε τον ανδρόνα δεν ήταν ε, πάντα μόνο θετικός. Υπήρχε αρκετή αντίδραση, μεγάλη αντίδραση για την ένταξη των γυναικών. Όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο τη δουλειά μας. Πρέπει να πω επίσης ότι η Επίτροπός μας που μπορεί σε κάποια θέματα να μην συμπίπτουμε στις απόψεις μας και εγώ έχω διαφορές απόψεων μαζί της, αν κάτι έχει ξεχωριστό, η Επίτροπος είναι ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Και έτσι λοιπόν πραγματικά την εκτιμούμε ιδιαίτερα ότι ήταν παρούσα εδώ και Κρίμα είναι ότι δεν προσήλθαν άλλοι ευρωβουλευτές εδώ. Η παρουσία της όμως είναι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε εδώ, ότι είναι ιδιαίτερα θετική εδώ. Επειδή εκείνη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι ευαισθητοποιημένη για να προασπιστεί τον ρόλο των γυναικών όσον αφορά την εργασία τους στον τομέα της αλίας. Και τώρα εν ώψη της μεταρρύθμισης στον τομέα της αλίας που πολλά πρόκειται να γίνουν, νομίζω όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή είναι η μάχη που δίνει, ο αγώνας που κάνει καθημερινά και με τα κονδύλια που ε, πολλές φορές σπανίζουν και με την ε, υποστήριξη που σπανίζει πολλές φορές και έναντι των κρατών μελών και θα έλεγα και από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αλλά να βασίζεστε μαζί μας στην υποστήριξή μας σε σχέση με το μέλλον και τις προσπάθειές σας. Ευχαριστώ όλους και λίγη εδώ αυτή η ακρόαση που είχαμε. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας κυρία Επίτροπε. Εδώ για την Επιτροπή Αλληλείας πρέπει να συνεχίσουμε με τα τελευταία θέματα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας μετά από την ακρόαση. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι τα διάφορα. Η κυρία Ντότς νομίζω ήθελε να θέσει κάποιο αίτημα ή κάποια ερώτηση. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Chair. Um, just... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώς μια σύντομη ερώτηση. Πρώτα απ' όλα με συγχωρείτε που δεν ήμουν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της ακρόασης, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή του ε, Προέδρου ε, διότι αυτό οφείλεται στο ότι επικαλύπτονται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Γεωργίας με τις Επιτροπής Αλίας. Αυτό συμβαίνει συνεχώς και αυτή είναι η εξήγησή μου, η δικαιολογία μου ε, για το ότι δεν ήμουν εδώ. Ως αναπληρώτρια μέλος θα ήθελα να παρακολουθώ στο δυνατόν περισσότερες ακροάσεις ε, είναι δυνατόν, αλλά τα σήμερα είχα μια άλλη συνεδρίαση. Θα ήθελα να θέσω μια απλή ερώτηση. Ε, έχουμε, θα έχουμε το Συμβούλιο Αλίας ε, το Δεκέμβριο και με εκπλήσει που οι ευρωβουλευτές δεν είχαν δυνατότητα να έχουν μια παρουσίαση για τις προτάσεις για το Συμβούλιο Αλίας και δεν είχαν την ε, δυνατότητα να συζητήσουν αυτές τις προτάσεις ε, ή να θέσουν ερωτήσεις στην Επιτροπή σε σχέση με τέτοιες προτάσεις. Διαρωτώ με, υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Εγώ έχω την εντύπωση και νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι αισθάνονται ότι είναι σημαντικό για ε, τις δημοκρατικά εκλεγμένους ε, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα θέματα αυτά. Ε, ξέρω βεβαίως ότι ε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, αλλά βεβαίως ε, η συζήτηση των θεμάτων θα ήταν ίσως πάρα πολύ σημαντική. Ίσως εγώ έλειπα. Ναι, και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση των τάξη και των ποσοστώσεων και για τις γενικές γραμμές αυτών που θα διαμορφώσουν τα τάξη και τα κβότα και τις ποσοστώσεις, τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Η πρόταση που θα υποβληθεί από την Επιτροπή θα συζητηθεί το Δεκέμβριο, δεν έχει συζητηθεί εδώ, όμως σε σχέση με μέχρι τη σημερινή ε, ημερομηνία δεν υπήρξε κάποιο αίτημα από κάποιον Οπότε, ανεξάρτητα από το τι θα μπορούσαμε εμείς να διακοπεί, ναι, μια παρουσίαση για την ανακοίνωση, μάλιστα. Επί της ανακοίνωσης ε, αυτής, σε σχέση με το τι θα συναποτελεί αυτή την πρόταση, αυτά θα είναι τα στοιχεία της πρότασης, έτσι. Για τη συγκεκριμένη πρόταση, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αν είχατε διατυπώσει αυτό το αίτημα πριν από αυτήν την τελευταία συνεδρίασή μας θα μπορούσαμε να το είχαμε λάβει υπόψη. Αλλά τώρα δεν βλέπω άλλη δυνατότητα, εκτός αν γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο της Επιτροπής μας. Αν μπορεί να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας, τότε και παραστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Δεν βλέπω άλλη δυνατότητα για να δοθεί κάποια απάντηση. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι μια έκτακτη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική μα επιτροπή στο Στρασβούργο, στην περίοδο συνόδου τη Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, ώστε να έρθει η Επιτροπή και να παρουσιάσει σε σχέση με την πρόταση που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών τα στοιχεία τη, αν συμφωνείτε. Sorry. Um, I, I was aware and I was Ναι, ναι, ε, ε, Θέλω τι ακριβεί προτάσει Είχα τη γενική παρουσίαση ε, πέρσι σε αυτήν την Επιτροπή έγινε μια παρουσίαση για τις πραγματικές προτάσεις της Επιτροπής και εγώ, ίσως και άλλοι στην Επιτροπή, είχαμε υποθέσει ότι αυτό θα γινόταν σήμερα. Μέχρι ότου είδα την ε, λεπτομερή ε, ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ε, δυνατότητα έκτακτης συνεδρίασης στο Στρασβούργο, διότι είναι ταυτόχρονα με το Συμβούλιο Υπουργών. Νομίζω ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ε, μια συζήτηση για τις, ε, πρότασεις, για τις προτάσεις του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου για την Αλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον του κλάδου. Η πρόταση για το κείμενο υφίσταται. Τώρα, δεν βλέπω κάποια δυνατότητα να υπάρξει μια επαφή με την Επιτροπή, μια συνεδρίαση με την Επιτροπή, εκτό αν είναι μια έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, όπου θα μπορούσε να προσέλθει και να ενημερώσει η Επιτροπή για αυτήν. Υπάρχει σε γραπτό κείμενο η πρόταση αυτή και οποιοδήποτε μπορεί να την έχει. Εγώ την έχω, την έχω αυτή την πρόταση όπως ε, αν θέλει κάποιος να την έχει και μπορεί να συζητήσει τώρα αυτή την πρόταση, ο μόνος τρόπος που μπορεί να γίνει είναι να έχουμε μια έκτακτη συνεδρία στο Στρασβούργο, όπως είπα. Αν συμφωνείτε σας. Αν, μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Bueno, Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα προσπαθήσω να το συζητήσω, να το συζητήσουμε στο Στρασβούργο. Το Συμβούλιο δεν, δεν θα ε, εμπλέκεται, έτσι δεν είναι. Μπορούμε να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Εν πάση περιπτώσει, η πρόταση υπάρχει και μπορούμε να την ε, έχουμε. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Θα δούμε με τους συντονιστές, θα δούμε τις ημερομηνίες και θα δούμε αν υπάρχει δυνατότητα να γίνει μια έκτακτη ξεχωριστή συνεδρίαση γι' αυτό στο Στρασβούργο. Λοιπόν, με αυτά περνάμε στο επόμενο σημείο στη μέση διάταξη, που είναι ανακοινώσει της Προέδρου σε σχέση με τις αποφάσεις ε, που υιοθετήθηκαν από τους συντονιστές. Διανεμήθηκε διανεμήθηκε ένα κείμενο με τις αποφάσεις ε, που ε, έλαβαν οι συντονιστές. Κυρία Ντότς, παρακαλώ. οι κυρίες παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με μένα το ίδιο συμβαίνει όπως με την συνάδελφο πιο πριν. Στην ακρόαση δεν μπόρεσα να συμμετάσχω, δυστυχώς επειδή προσωπικά δεν μπορώ να διχαστώ σε δύο, δεν μπορώ να είμαι σε ένα σημείο και σε ένα άλλο δυσυπόστατα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα της παρέμβασής μου, θα ήθελα να σας παρακαλέσω στα πρακτικά να καταχωρηθεί ότι οι ευρωβουλευτές, τα μέλη, θα ζητηθεί, θα παρακληθεί στις κυβερνήσεις τους να απευθύνουν μια επιστολή στους υπουργούς αλίας, αρμόδιους υπουργούς αλίας των κυβερνήσεών τους, όπως το είχαμε συζητήσει χθε, δεν είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά. Θα ήμουν ευγνώμων αν θα τα κοτοχαρούσαμε στα πρακτικά. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θα προσκληθούν θα προσκληθούν να συντάξουν αντίστοιχε επιστολέ που θα απευθύνουν στου αρμόδιου ε, εθνικού υπουργού αλεία. Αυτό είχα ζητήσει και παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ. Πολύ καλά θα καταχωρηθεί στα πρακτικά αφού το αυτό επιθυμείτε. Αλλά εδώ δεν είναι κάτι που είναι μια συμφωνία που απαιτεί ε, το υποχρεωτική ε, συμμόρφωση. Αν θέλετε λοιπόν εσείς αυτό να καταχωρηθεί στα πρακτικά, πολύ καλά. Δηλαδή οι βουλευτές να απευθύνουν μια επιστολή στους υπουργούς των κρατών μελών των κυβερνήσεων να παροτρύνουν να ληφθεί μια απόφαση για το θέμα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Εντάξει, δεν ξέρω ποια επίπτωση θα είχε μια τέτοια επιστολή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια και δεν είναι μια υποχρεωτική μορφή συμφωνίας, αλλά είναι κάτι που είναι μια σύσταση. Είναι μια σύσταση. Μπορούμε να το πούμε, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι, δεν υποχρεωμένος κανείς να συμμορφωθεί. Ούτε και αυτό όμως είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο να θέτει προβλήματα. Μια και δεν υπάρχει άλλος από εσά ε, εδώ, το θέμα, για το θέμα αυτό μπορεί έτσι να ρυθμιστεί. Περνάμε στη συμμετοχή τώρα στις ακροάσεις. Όλοι έχουμε αρκετές κοινοβουλευτικές επιτροπές, αυτό είναι δεδομένο θέμα. Κάθε ένας έχει τις προτεραιότητες και τις αντιλημμένες υποχρεώσεις του. Και είναι και καλό αυτό. Είναι θέμα προτεραιοτήτων όμως, γιατί αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα. Περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Η ημερομηνία διεξαγωγής προσεχού συνεδρίασης θα γίνει καταρχήν, εκτός αν υπάρξουν, υπάρξει κάποια έκτακτη συνεδρίαση, θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου και στις 26 Ιανουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες οι συνεδριάσεις μας. Να υπενθυμίσω εκ νέου ότι ε, την, ε, ε, στις 7 Δεκεμβρίου στις 5 η ώρα θα έχουμε ένα κόκτελ που θα παραθέσει η Επιτροπή μας και προς τους διερμηνείς και όλους. Να υπενθυμίσω, 7 Δεκεμβρίου είναι αυτή η ημερομηνία, εντάξει. Και με όλα αυτά σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας εδώ, για τη δουλειά σας. Γεια σας, καλό βράδυ.